κανονισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη κάποια επιχειρησιακά ζητήματα. Εδώ δεν καθορίζονται τα όρια της συγχωρήπανσης ε, γιατί υπάρχει άλλη οδηγία η οποία ασχολείται με τα ε, όρια του, του, του θορύβου κτλ. Ε, επομένως εδώ δεν μπορούμε να καθορίσουμε ας πούμε δεσιμπέλ στο κείμενο αυτό. Ε, και επομένως ε, απλώς ε, μπορούμε να αναφέρουμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρησιακές αποφάσεις όσον αφορά την μείωση του, της ηχορύπανσης. Αυτό που θέλουμε εδώ είναι να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης της ηχορύπανσης έχουν ξεπεραστεί λόγω και των τεχνολογικών πρόοδων ε, τα όσα ανεφέρονται στην προηγούμενη οδηγία η οποία είναι δεκαετίας πλέον ε, και επομένως ε, κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Υπάρχει και μία τροπολογία η οποία δεν θα αρέσει στην Κομισιόν και εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να είναι κανονισμός αλλά οδηγία και αυτό ε, δημιουργεί συζητήσεις ε, με την ε, Κομισιόν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα εξειδικευμένα προβλήματα στα αεροδρόμια όσον αφορά το επίπεδο θορύβου. Πήγαμε σε πολλά αεροδρόμια ε, τα αεροδρόμια της Ευρώπης ε, διαφέρουν και όσον αφορά την κατάσταση και όσον αφορά το μέγεθος και όσον αφορά ε, την, το βάρος της κυκλοφορίας κτλ. νομίζω ότι μπορούμε να προτείνουμε την ε, την μείωση ε, κάποιων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αλλά ξέρετε ε, σε μερικές περιπτώσεις αυτό μπορεί να αποτελέσει να έχει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα όσον αφορά ας πούμε τις νυχτερινές πτήσεις υπάρχουν κάποια αεροδρόμια στα οποία μπορούν κάλλιστα να γίνονται νυχτερινές πτήσεις ενώ σε άλλα δεν είναι καθόλου εύκολο θα πρέπει λοιπόν η ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικέ συνθήκες και βεβαίω είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις ιδέες που θα μπορούσαν να υποβληθούν ε, για το θέμα αυτό. Κάτι άλλο τώρα. Η δυνατότητα ε, νυχτερινών τερματικών σταθμών. Προτείνεται η ένδειξη νυχτερινός τερματικός σταθμός. Κοιτάξτε, εμείς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με απλό ταχυδρομείο και μέσω της Επιτροπής Αναφορών λάβαμε ε, σωρία παραπόνων ε, όπου αναφέρεται σαν κύριο πρόβλημα ε, οι νυχτερινές πτήσεις. Ε, υπάρχουν ας πούμε κάποιες πτήσεις οι οποίες είναι εμπορικές και οι οποίες ε, ε, είναι απαραίτητες. Εμείς δεν λέμε ότι θα πρέπει να σταματήσει ή να πληγεί η οικονομική δραστηριότητα. Απλώς θα πρέπει αυτή η οικονομική δραστηριότητα να ε, ε, αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο, να τη διαχειριστούμε με πιο βιώσιμο τρόπο και με πιο σωστό και για το περιβάλλον και για τους γείτονες που υφίστανται πολλών ειδών ρυπάνσης. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ήθελα να πω ε, που αφορά την χωροταξία. Βεβαίως αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως μπορούμε να κάνουμε και κατά αυτή την έννοια κάποιες συστάσεις. Ε, να στραφούμε λοιπόν προς τους εμπλεκόμενους φορείς, να στραφούμε ε, προς τις τοπικές αρχές για να κάνουμε κάποιες συστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή θα πρέπει η διαχείριση του αεροδρομίου, του όποιου αεροδρομίου, να λαμβάνει υπόψη της ε, και τις ε, μελλοντικές επεκτάσεις του αεροδρομίου αυτού και να πούμε εξ αρχής ε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, σε ποιες περιοχές δεν μπορεί να επεκταθεί κτλ. Αυτό καλό είναι να το ξέρουμε εξ αρχής, να δούμε επίσης τι μπορεί να γίνει κοντά στο αεροδρόμιο. Ε, ας πούμε πολλές φορές ε, δίνεται άδεια για την λειτουργία ενός αεροδρομίου ενώ πολύ κοντά ε, έχουν δοθεί άδειες οικιστικές και στο τέλος οι γείτονες δεν μπορούν να κοιμηθούν. Είπα λοιπόν ότι θα πρέπει και να ξεκαθαρίσουμε και την έννοια των ενδιαφερομένων φορέων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θίγονται άμεσα ε, και επίσης ε, στο κείμενο δεν γίνεται αναφορά στους τοπικούς φορείς. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να θεωρηθούν εμπλεκόμενοι φορείς ε, και επομένως να αναφερθούν και στο κείμενο. Θα πρέπει να προβλέπονται διαβουλεύσεις, θα πρέπει να προβλέπεται διαδικασία σφιγμομέτρησης, λήψης ε, των αποφάσεων και από εκεί. Ε, πρέπει να πούμε ότι ε, πολύ συχνά η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πολύ καλές γνώσεις τεχνικές και τεχνολογικές και επομένως μπορούμε να, και σε συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς να βρούμε σωστές ισορροπημένες λύσεις. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν ε, στην οικονομική δραστηριότητα αλλά και οι φυστάμενοι ε, της ζημίας της δραστηριότητας αυτής ε, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διαβούλευσης. Αυτή τη στιγμή είναι πολλοί οι θυγόμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τριβές ή αντιμετωπίζουν διαμάχες πολύ δύσκολο να επιληθούν. Εμείς ε, δίνουμε τη δυνατότητα στους φυγόμενους ε, ε, να λάβουν τα μέτρα τα οποία προβλέπονται. Όταν υπάρχει κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε με την Κομισιόν, γιατί πρέπει να ακούσουμε και τους ενδιαφερόμενους, που λένε ότι είναι λίγο υπερβολικά αυτά τα οποία προβλέπονται Βλέπετε από την Κομισιόν όταν υπάρχει ένας λειτουργικός ε, περιορισμός που επιβάλλεται ε, λέγονται κάποια πράγματα αλλά δεν λέει τίποτα ένας λειτουργικός ε, περιορισμός που πρέπει να οριστεί δεν ορίζεται και οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν ένσταση ώστε να γίνει αυτό. Είναι δικατευθυντικό, αμφίδρομο όλο αυτό και πρέπει να είναι ξεκάθαρο. και πρέπει να υπάρξει μια εξισορρόπηση σε αυτή την παρέμβαση της Κομισιόν και να μπορούν και οι ενδιαφερόμενοι να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει, αν δεν έχει προβεί ενέργειες, στις δέουσες ενέργειες. Για να μην μακρηγορήσω ιδιαίτερα με το κείμενο που είχαμε και βέβαια με τις δυνατότητες που έχουμε ως Κοινοβούλιο, θελού, θελήσαμε να υπάρχει ενημέρωση, να υπάρχει διαφάνεια για όλη την ε, διαδικασία, να δίνονται οι απαραίτητε πληροφορίε στου ενδιαφερομένου, γιατί να αποκρύπτονται δεν έχει καμία, κανένα απολύτω ε, ε, νόημα. Διότι σε κάποιε περιοχέ κοντά σε αερολιμένε βλέπουμε να αποκρύπτονται κάποιε πληροφορίε. και κάποιες φορές υπάρχουν κάποια ε, αλλαγές δρομολογίων που δεν δικαιολογούνται από κάποιο έκτακτο γεγονός, ε, ούτε κάποιο γεγονός που έχει να κάνει με τον καιρό, ούτε τίποτε άλλο. Επίσης, ένας πολύ σημαντικός ε, παράγοντας είναι ο περιβαλλοντικός και ο παράγοντας της δημόσιας υγείας, της υγείας ε, των ανθρώπων, της ανθρώπινης υγείας. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, αν θέλουμε να είμαστε ισορροπημένοι στην προσέγγισή μας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία. Επίσης, ε, υπάρχει και η ισορροπία στον έλεγχο των εξουσιών τη Κομισιόν. Αυτοί είναι τέσσερις άξονες. Εκεί πάνω βασίζονται οι τροπολογίε μα. Έτσι, πιστεύω ότι παρότι εκπονούμε μία γνωμοδότηση, θα αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά αυτή την έκθεση, που δεν είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε ελαφρά, είναι πολύ σοβαρό το θέμα παραμένω στη διάθεσή σας, ε, είτε αν έχετε κάποια απορία, είτε για να συζητήσουμε ορισμένα σημεία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την πολύ λεπτομερή παρουσίαση της προβληματικής που είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδης Τζακλίν Φώστερ, μόνο αυτή έχει ζητήσει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ο κύριος Νέλχαρτ θέλει να παρέμβει. Άλλος, Καρλ Χάιντς Φλόρεντς, Ζακλίν Φώστερ, Σνέλχαρτ, Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ο Κούρτο Χόλσκι έλεγε ότι ο θόρυβος είναι ο θόρυβος που κάνουν οι άλλοι. Είμαστε μέλη της Επιτροπής Υγείας και άρα πρέπει να δούμε και πώς επηρεάζει ο θόρυβος την υγεία. Ξέρουμε από πόσα δεσιμπελ και πάνω είναι επικίνδυνος ο θόρυβος. Βέβαια, η ευαισθησία στο θόρυβο είναι υποκειμενικό. Ε, μετράται υποκειμενικά. γνωρίζουμε ότι όσο περισσότερο εκτίθεται ο άνθρωπος ε, στο θόρυβο, τόσο πιο ευαίσθητος γίνεται και τόσο πιο ε, μεγάλο άγχος και στρες αναπτύσσει και για τον πόνο και για το θόρυβο δεν υπάρχει συνήθεια, δεν συνηθίζεται ο θόρυβος ή ο πόνος. Και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες σε σχέση με την χορύπανση. Δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε στον κανονισμό υπόψη μόνο ε, τις οικονομικές παραμέτρους στις αερομεταφορές. Είναι μείζον θέμα η δημοσιογεία και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει επίσης ε, να λαμβάνουν υπόψη και τις ιδιαιτερότητες που έχει η τοποθεσία ενός αερολιμένου. Και οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται επί τόπου σε συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό. διότι μόνο στο τοπικό επίπεδο μπορούν να βρίσκονται εξατομικευμένες αποφάσεις και να λαμβάνονται τέλος πάντων οι αποφάσεις. Και ε, εγώ υποστηρίζω την ε, προσέγγιση ε, του εισηγητή Περέλο όσον αφορά το άρθρο 10 ε, που προστατεύει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί με συμμετοχή των πολιτών. Αλλά δεν θέλουμε η Επιτροπή να μπορεί να απορρίψει μια απόφαση που έχει ληφθεί με συμμετοχή των πολιτών. Θα πρέπει να τηρούνται οι υποσχέσεις που γίνονται και θα πρέπει να υπάρχει ένα αξιόπιστο πλαίσιο. Κανένα αεροδρόμιο δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Συνδέεται με το σύνολο του ε, δικτύου των αερομεταφορών. Πριν δύο χρόνια είχαμε τον έφος στάχτης πάνω από την Ευρώπη και είδαμε ότι πολλές επιχειρήσεις ε, δεν μπορούσαν να παράγουν διότι δεν ε, είχαν αρκετές ε, ύλες αποθηκευμένες. Αν δεν υπάρχει εργασία δεν υπάρχει και πληρωμή μισθών. Θα πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά και η συνεργασία είναι πολύ σημαντική. Η διαμεσολάβηση που έχει συμπεριλάβει ο εισηγητής στην εκθεσή του είναι επίσης σημαντικό στοιχείο. Και δεν μιλάμε για το, τα αεροδρόμια μιας χώρας, ε, η Ευρώπη έχει ε, ε, διασυνδέσεις με όλο τον κόσμο. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και τα συμφέροντα όσον αφορά την υγεία και τα οικονομικά. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της ε, παράτασης των προθεσμιών. Εάν δηλαδή έχουμε παράταση ένα μήνα αντί για τρεις, ε, θα πρέπει να δούμε ε, ποιες είναι οι συνέπειες. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο Περέλο τι εννοεί όταν μιλάει για αεροσταθμό νυχτερινών πτήσεων. και πώς ε, θα γίνει η μεταφορά μετά των επιβατών από εκεί. Από το δρόμο θα γίνει. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε πολλά με μια τέτοια πρόταση. Ε, υπάρχει πρόταση για υποβάθμιση του κανονισμού σε οδηγία. Για μένα πρόκειται για υποβάθμιση. Ε, εγώ θα ήθελα να επιλέξουμε το μέσο που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε καλύτερα το στόχο μας. Και σε έναν κανονισμό μπορούμε να επιτρέψουμε περιθώριο για εθνικές αποφάσεις και για την επικουρικότητα. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν. Δεν είμαι ειδική στα θέματα αυτά, αλλά η Κομισιόν έχει ασχοληθεί εντατικά με το θέμα. Έχουν εξεταστεί όλες οι ευφυείς και καλές λύσεις εδώ. Διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ένα αποτελεσματικό δίκτυο. Και να μην κοιτάμε το κέρδος μόνο κάθε μεμονωμένο αεροδρομίου. Θα πρέπει να έχουμε οργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ε, μεταφορά των επιβατών και των αγαθών ε, στον προορισμό τους. Επίσης ε, έχουμε εδώ το παράδοξο ότι από τη μία ο πολιτισμός ε, οδηγεί σε νέες πηγές θορύβου, αλλά οδηγεί και σε αυξημένη ανάγκη για ανάπαυση και ησυχία. Θέλουμε όλοι, για παράδειγμα, να πηγαίνουμε γρήγορα και φθηνά διακοπές. Τι είναι δυνατόν λοιπόν και πώς αξίζει τελικά η ανάπτυξή μας. Πόσες μεταφορές θέλουμε και πόσες χρειαζόμαστε και πόσο θόρυβο μπορούμε να αντέξουμε. Αυτό είναι το θέμα που θα πρέπει να εξετάσουμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε το θέμα του θορύβου ως προς ε, τις ε, συνέπειες του στην υγεία στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέα Τσανώνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του. Ως σκιώδης εισηγητής από την ομάδα Άλντε θα κάνω κάποια γενικά σχόλια διότι δεν έχω μελετήσει και τις το τροπολογιστή του κυρίου Περέλου. Όπως όμως ε, πολύ σωστά υπογράμμισε ο εισηγητής, η χορύπανση ιδίω των νυχτωρινών πτήσεων επηρεάζει αρνητικά το φυτικό επίπεδο τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων πολιτών που ζουν κοντά σε αεροδρόμια και οι οποίοι, όπως ε, υπενθυμίζω εισηγητή, ε, ουσιαστικά υποβάλλονται σε τριπλή ρήπανση. Χορύπανση, ατμοσφαιρική ρήπανση και χημική ρήπανση. Ιδίω ο νυχτερινό ε, θόρυβο, όπω αναγνωρίζουν διεθνεί επιστημονικέ μελέτε, προκαλεί σοβαρέ βλάβε για την υγεία. Οι περισσότεροι βέβαια άνθρωποι που ταξιδεύουν θέλουν να διατηρήσουν την, ε, τις πολυάριθμες επιλογές ε, που έχουν στη θέση τους. Και πολλές φορές η αεροπορική κυκλοφορία είναι και ένας παράγοντας τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης. Πώς λοιπόν θα συνδυάσουμε αυτές τις δύο απαιτήσει, αυτούς τους δύο στόχους λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι είμαστε η Επιτροπή που είναι αρμόδια για το περιβάλλον, αλλά και τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών. Προτεραιότητα για μα λοιπόν έχουν οι καταναλωτέ. Η αρμόδια καθήλυν Επιτροπή, η Επιτροπή Μεταφορών, θα εξετάσει και τη δική μα τοποθέτηση. Επομένως, υποστηρίζω πλήρως τον εισηγητή, ο οποίος προσπαθεί να βελτιώσει ε, την ε, προστασία των πολιτών όταν αυτοί εκτίθενται σε αυτού του είδους την ηχορύπενση και μιλά για μια ισορροπημένη προσέγγιση δεν είναι όμως εξίσου πιστική η θέση του εισηγητή εκεί όπου θεωρεί ότι μια οδηγία ε, θα ήταν καλύτερο εργαλείο έτσι ώστε να επιτύχουμε καλύτερη προστασία των πολιτών που υφίστανται την ηχορύπανση. Στόχος της ε, πρότασης ε, είναι να οριστεί μέθοδος ε, καθορισμού της ηχορύπανσης. Εδώ όμως δεν επισέρχεται εις τις λεπτομέρειες οι οποίες δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με την Οδηγία 49 ακολουθούνται τα εθνικά σχέδια δράσης για τα όρια της ηχορύπανσης. Φαίνεται λοιπόν ε, να είναι πιο πιστική η επιλογή της Κομισιόν, ε, δηλαδή οδηγία, η οποία, κανονισμός συγγνώμη, ο οποίος θα εφαρμόζεται ε, ανάμεσα, άμεσα και που θα μπορεί να εναρμονίσει τις δραστηριότητες όλων των πολιτών. Βεβαίως ε, είναι σημαντικό ο εκπρόσωπος της Επιτροπής να πάρει το λόγο έτσι ώστε να μας πει την άποψή του για αυτό το σημαντικό θέμα. Ε, επίσης και άλλα σημαντικά θέματα εισάγει η πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ας πούμε πιο αυστηρή ε, ε, πιο αυστηρούς ορισμούς και περιορισμούς όσον αφορά τα ειδικά ε, αεροπλάνα τα οποία δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στους γείτονες. Επίσης, συμμεριζόμαστε την πρόταση για ύπαρξη σαφών κανόνων σε σχέση με το ποιοι είναι οι φορείς οι οποίοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην διαβούλευση για την ηχορύπανση. Επίσης, ε, η υποχρέωση των ε, κρατών μελών ε, για τακτική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Θα υποβάλλουμε λοιπόν και κάποιες τροπολογίες οι οποίες κατά την άποψή μας συμπληρώνουν την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζανώνη. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στη συνάδελφο Γιανακουδάκη. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Μου άρεσε η προσέγγιση του. Πρώτα υγεία είναι μια πολύ σωστή προσέγγιση. Σίγουρα πρέπει να βλέπουμε και πού βρίσκονται τα αεροδρόμια. Είναι αστική περιοχή, είναι αγροτική περιοχή, πώς επηρεάζεται η περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Αλλά σε αντίθεση με τους άλλους δύο σκιώδεις δεν, με, ε, δεν μου προκαλεί ιδιαίτερο πρόβλημα το αν θα είναι οδηγία αντί κανονισμός. Εγώ δεν βλέπω έτσι να υποβαθμίζεται, αλλά να αναβαθμίζεται η έκθεση. Γιατί είναι καλό να υποστηρίζεται και από την τοπική κοινωνία. Θέλω να δω λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η επιχειρηματολογία αν είναι τοπικό το αεροδρόμιο, πρέπει να συμμετέχει ο τοπικό κόσμο, η τοπική κοινωνία. Θα πρέπει όμω να είμαστε και ευαίσθητα απέναντι στη βιομηχανία που προσφέρει θέσει εργασία, προσφέρει δουλειέ στου ανθρώπου αυτού. Και νομίζω ότι η βιομηχανία κάνει πολλά για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συγχώρυπανσης με τα αεροσκάφη του κεφαλαίου 4, θα γίνει καλύτερα να έχουν και το κεφάλαιο 5 που βοηθά να υπάρχει, μάλλον να ενισχύει τις προσπάθειες για μεγαλύτερη χωμόνος, όπως προσπάθειες που γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, οικονομική ε, ανάπτυξη της τα κτλ. Δεν μπορούμε δηλαδή να παραγνωρίζουμε και το θετικό σκέλος. Σίγουρα η υγεία είναι πρώτο μας μέλημα βέβαια. Σε ό,τι αφορά τώρα τις νυχτερινές πτήσεις ή τους νυχτερινούς θερματικούς σταθμούς, δεν είμαι 100% σίγουρη για το πώς αυτό θα λειτουργήσει και αν μπορεί να λειτουργήσει διότι ο νυχτερινός θόρυβος ε, είναι το ίδιο κακός ε, με τον ημερήσιο αν σου διακόπτει τον ύπνο. Δεν ξέρω αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επηρεάσει τις αποφάσεις των τοπικών αρχών ε, για τον προγραμματισμό. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποτελεί αρμοδέ των τοπικών αρχών. Εγώ θα έλεγα ευελιξία. Πρέπει να δοθεί ευελιξία στα κράτη-μέλη για να κάνουν αυτά που καλύτερα ταιριάζουν στο κάθε κράτος. Μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των τοπικών αρχών. Αυτά θα ήταν προτεραιότητές μου. Έτσι τα συνοψίζω. Πάντως θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βίλς. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια μέρα ο άνθρωπος θα πρέπει να καταπολεμεί το θόρυβο σαν την ε, χολέρα. Ε, αυτό είπε ο Ρόμπερ Κόφ πριν 100 ε, χρόνια και φτάσαμε στην εποχή αυτή. Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε κάτι, αλλά διαπιστώνω ότι το σχέδιο κανονισμού της Κομισιόν δεν είναι κατάλληλο για να μειώσει τον θόρυβο στα, στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής ο κανονισμός αυτός λόγω της μονομερούς κατεύθυνσής του ε, ασχολείται κυρίως με την αύξηση της, ε, του, του δυναμικού των ευρωπαϊκών αεροδρομίων και γι' αυτό θα πρέπει να ε, τον απορρίψουμε. Η καταπολέμηση του θορύβου παίζει δευτερεύοντα ρόλο στον κανονισμό αυτό. Το τι ενδιαφέρει την Κομισιόν φαίνεται στο εκτιμώντας εννέα ότι τα μέτρα για περιορισμό του θορύβου θα πρέπει να μπορούν να αναβληθούν ε, για να αποφύγουμε ανεπιθύμητες συνέπειες ε, στο δυναμικό των αεροδρομίων, ε, στην ασφάλεια κλπ. Εμείς θέλουμε περιορισμό της ε, λειτουργίας, ε, το οποίο σημαίνει ε, απαγόρευση των νυχτερινών πτήσεων. Η Κομισιόν θέλει τη δυνατότητα αναβολής της απαγόρευσης, εάν το θέλει, ένα κράτος μέλος ή και από μόνη της, αν το επιθυμεί. Οι πολίτες που ζουν κάτω από αεροδιαδρόμους διαμαρτύρονται, δεν μπορούν να δεχτούν άλλο αυτή την κατάσταση στη Φραγκφούρτη και στο Βερολίνο δεν ζητήθηκε από τις αρχές απαγόρευση των νυχτερινών πτήσεων, αλλά ε, ε, δόθηκε εντολή από ε, δικαστή. Μπόρεσαν έτσι οι άνθρωποι τουλάχιστον εν μέρη να πετύχουν αυτό που ήθελαν. Εάν όμως τώρα η Κομισιόν άρει τέτοιες απαγορεύσεις, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι υπερβολικό. Ε, ο κανονισμός αυτός φέρει την υπογραφή των ε, αεροπορικών εταιριών και φαίνεται ότι αυτές είναι πιο σημαντικές για την Κομισιόν από ότι η υγεία και ε, η ευημερία των ανθρώπων. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία. Το σχέδιο του εισηγητή πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν προχωράει όμως αρκετά. Όπως ήδη έγινε σαφές, ε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ε, πολύ λίγο τα οικολογικά θέματα και περισσότερα τα θέματα κόστους όφελους. Ε, με τη θέση του εισηγητή ότι δεν είναι αναλογικό μέτρο ε, να επιλέξουμε οδηγία αντί για όπως προτείνει η Κομισιόν. Ωστόσο, τα νυχτερινά ε, αεροδρόμια ε, πιστεύω ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Βλέπω επικριτικά την ιδέα αυτή. Δεν ε, πρόκειται να συμβάλλουν στη μείωση του θορύβου και των συνεπειών του στις στην υγεία των πολιτών. Του αντίον πιστεύουμε ότι ανοίγει την πόρτα για περαιτέρω αρνητική, αρνητικές επιπτώσεις. είναι απαραίτητη ε, η καλύτερη συνδρομική διασύνδεση σε μικρές αποστάσεις, ε, διότι η μεταφορά αγαθών με τα αεροπλάνα δεν είναι ούτε οικονομική ούτε οικολογική. Κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Πολύ ενδιαφέρουσα πρότασή του. Νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι της Επιτροπής έχουν θέσει κέρια ζητήματα εγώ στηρίζω τον εισηγητή και μάλιστα το συζητήσαμε στην Επιτροπή Μεταφορών στο κατά πόσον θα πρέπει να πρόκειται για κανονισμό ή οδηγία. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα επικουρικότητας σε σχέση με αυτή την έκθεση. Μας ανησυχεί λοιπόν το να μετακινηθεί, να γίνει από οδηγία κανονισμός γιατί θα μπορούσε να υποβαθμιστεί ε, το τοπικό επίπεδο και δεν θα θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο, περισσότεροι από εμάς. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, τον κατεξουσιοδότηση πράξεων και πάλι εδώ ορισμένοι από εμάς ανησυχούμε με το άρθρο 10. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άποψή μου θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις κατεξουσιοδότηση πράξη. μόνο για τεχνικές επικαιροποίησεις. Άρα εδώ βάζουμε ερωτηματικό. Για άλλα θέματα τώρα παραδείγματο χάρη εύρο τοπική αντιπροσώπευση κτλ. Είναι ε, θεμητό να υπάρχει εκπροσώπηση και ίσως και άλλοι θα πρέπει να ενημερώνονται, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί υπάρχουν πολύ ενδιαφερόμενοι, πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση υπάρχουν ομάδες πίεσης που δεν λογοδοτούν σε κανέναν και όσοι ενδιαφέρονται ε, με αυτά, ε, για αυτά τα θέματα θα πρέπει να λογοδοτούν και να είναι υπόλογοι ε, όσοι συμμετέχουν ιδίω και σε κάποιες ομάδες γιατί αλλιώς δεν θα έχουν καμιά ευθύνη, δεν θα δίνουν λόγο σε κανέναν πρέπει λίγο να το σκεφτούμε Σε ό,τι αφορά τώρα το χωροτεξικό σχεδιασμό, το σχεδιασμό της χρήσης της γης είναι πολύ σημαντικό θέμα. Οι τοπικές αρχές στην Ευρώπη αλλά και παντού στον κόσμο Νομίζω ότι πολλές φορές ε, πήραν αποφάσεις για την έγερση ιδιωτικών κατοικιών πολύ κοντά σε αεροδρόμια και αυτό δεν έχει βοηθήσει καθόλου την ε, κατάσταση. Σίγουρα υπάρχει και πρόβλημα με την χωρητικότητα σε μεγάλους κόμβους. Όλα αυτά πρέπει να λυθούν υπόψη. Ολοκληρώνοντα, το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει τρόπου με του οποίου θα μπορούσαν να μετριαστούν οι δυσκολίε στα αεροδρόμια. Αν δει κανεί τι τεχνικέ πτυχέ, η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο. Εμείς στηρίζουμε την κοινή τεχνολογική ε, πρωτοβουλία Clean Sky, ε, τα αεροσκάφη δεύτερης γενιάς, 1,4 δις ευρώ ε, σε αυτό το σχέδιο, που είναι μια σύμπραξη δημοσιοδιωτικού τομέα. Πρέπει να δούμε και πάλι αν μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει για τη μετρίαση των λειτουργικών, επιχειρησιακών πιέσεων. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να λέγονται. Γενικά εμείς Νομίζω ότι θα δραματίζουμε ένα θετικό ρόλο για να προωθήσουμε αυτή την εξισορροπημένη προσέγγιση. Θα υπάρχουν πιέσεις, παρά το ότι εμείς θα προσπαθούμε να πιέζουμε για τις ε, ε, αρχές της ΔΟΠΑ. Τώρα αυτή είναι η χτερινή τερματική σταθμή. Παντού μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιο σταθμό, αλλά ουσιαστικά μεταθέτουμε το πρόβλημα. Το πηγαίνουμε από μια περιοχή σε μια άλλη. Και για σκεφτείτε ότι πολλές φορές ε, τα επιβατικά αεροσκάφη περιλαμβάνουν και πενταφέρουν και το μεγαλύτερο βάρος, ε, τα περισσότερα εμπορεύματα, αν σκεφτείτε ότι όλοι μας κυκλοφορούμε με ένα λάπτοπ ή οτιδήποτε άλλο και ανεβαίνουν στα αεροπλάνα. Νομίζω όμω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά το τι κάνουμε και εμεί εδώ στο Κοινοβούλιο με τι εκθέσει που εκπονούμε. Χωστ Σνέλχαρτ. Ε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα που συζητάμε. Και θα ήθελα να τονίσω ε, μία λέξη στον τίτλο ε, αυτού του θέματος. Ε, λέει «Ισορροπημένη προσέγγιση». Ξέρουμε ότι ο καθένας θα έχει αντίρρηση όσον αφορά το θόρυβο, είναι επιβάρυνση ο θόρυβος, επιδεινώνει την υγεία. Αλλά αν σκεφτούμε πόσο πιο ήσυχα έχουν γίνει τα αεροπλάνα τα τελευταία χρόνια, ε, πόσα μέτρα έχουμε ε, λάβει κατά του θορύβου στα αεροδρόμια, πολλά έχουν γίνει. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τελείως την οικονομική πτυχή, διότι δεν έχει νόημα αν δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αγαθά, κάτι που χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτή την εποχή. Να πούμε ότι αν δεν θέλουμε θόρυβο από τα αεροπλάνα, άρα δεν έχουμε πτήσεις. Αυτό δεν θα μας βοηθήσει πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. το, ε, οι αερομεταφορές είναι μια οικονομική πτυχή ε, ε, η χολέρα δεν είχε τίποτα θετικό δεν, πιστεύω λοιπόν ότι είναι τελείως λανθασμένη η σύγκρισή σας θα ήθελα να συζητάμε πιο λογικά το θέμα αυτό φυσικά οι άνθρωποι που ζουν κοντά στα αεροδρόμια, επιβαρύνονται. Εκτός, ε, παρατήρηση, ε, εκτός μικροφώνου μια παρατήρηση. Ε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακή η ιδέα με τα νυχτερινά αεροδρόμια. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης διότι έτσι μπορούμε να διατηρήσουμε την οικονομική πτυχή χωρίς να επιβαρύνονται με θόρυβο οι πολίτες. Και χρειαζόμαστε περισσότερους σιδηροδρόμους. Ξέρουμε όμως ότι ε, οι σιδηρόδρομοι σε κάποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φτάσει στα όρια του δυναμικού τους. Και άλλωστε και το τρένο το ακούει κανείς και αυτός είναι θόρυβος. Ούτε τα τρένα είναι ε, ε, τελείως ήσυχα. Χρειαζόμαστε κανονισμό διότι πρέπει να σκεφτούμε με ευρωπαϊκό τρόπο και όχι περιφερειακό. Πρέπει να συμφωνούμε όσον αφορά τους στόχους και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Καλ Χάινς Φλόρενς. Καταρχήν ε, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Κλάς. Η επικουρικότητα θα πρέπει να παραμένει σημαντική πτυχή. Υπάρχουν όμως και κάποιοι τομεί, όπου η επικουρικότητα για μένα ε, είναι υπερβολική. Εγώ μένω κοντά στο αεροδρόμιο του ε, Düsseldorf και όταν ε, βλέπω τι επιρροή έχει ο γερμανικός και αγγλικός στρατός όσον αφορά τις αφήξεις και αναχωρήσεις, και μάλιστα εάν ε, στο Μάστριχτ ε, πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο ύψος στα αεροπλάνα θα πρέπει να γίνουν τελείω διαφορετικά τα πράγματα στο Ντίσσελντορφ. Ε, μπορώ να φανταστώ ε, μια ε, διαμεσολάβηση της Κομισιόν, όχι όμως να λαμβάνει μόνο τις αποφάσεις. Ε, χθες συζητήσαμε το θέμα του θορύβου στα αυτοκίνητα. Και κάποιος που δεν θέλει θόρυβο, δεν θέλει αυτοκίνητα. Εγώ είμαι παθιασμένος οδηγός αυτοκινήτου και θέλω να, να συνεχίσω να οδηγώ αυτοκίνητο. Οι ε, αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να βρουν πιο σύγχρονα αυτοκίνητα. Πάντως γενικά βρίσκω πολύ καλή την πρόταση. Ευχαριστώ Καρφάνς Φλόρενς. Έτσι ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών συζητήσαμε ευρέω και εκεί είναι σαφές ότι ο θόρυβος ε, δεν είναι μόνο πρόβλημα στις αερομεταφορές ε, και στα αυτοκίνητα, αλλά και ε, στους σιδηροδρόμους. Θα πρέπει λοιπόν ω Επιτροπή Περιβάλλοντος να εξετάσουμε τις επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία όσον αφορά διάφορες πηγές θορύβου. και μήπως ε, εξάγουμε θόρυβο από νυχτερινές πτήσεις σε άλλα μέρη του κόσμου. Ε, θα πρέπει και αυτό να το έχουμε κατά νου αν απαγορεύσουμε τις ε, νυχτερινές πτήσεις. Με απαγόρευση άλλωστε δεν θα πετύχουμε τίποτα, θα πρέπει να έχουμε τεχνικές προόδους. Υπάρχει πάντως περιθώριο να περιοριστεί ο θόρυβος. Την Κυριακή θα γίνει ψηφοφορία στο Μόναχο. Ε, τρίτος σιδηροδρομικός σταθμός δεν θα ε, χτιστεί και ο βασικός λόγος είναι ο θόρυβος. Και άλλωστε όταν θα έχουμε ολοκληρώσει την ημερήσια διάταξη ε, θα μπουν όλοι οι συνάδελφοι στα αεροπλάνα τους και θα πάνε στις πατρίδες τους. Ε, ε, χρειάζεται λοιπόν συζήτηση στο θέμα αυτό. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις. Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρατηρή σας. Πραγματικά βρίσκονται στο επίκεντρο. Το ότι πρέπει δηλαδή να καταλήξουμε σε μια σωστή ισορροπία που θα λαμβάνει υπόψη ε, τις ανάγκες αλλά και τις προσδοκίες των συμπολιτών. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή Αντρές Περέγιο και για την έκθεσή του και για τις πολλές ε, και ενδιαφέρουσες ιδέες που περιέχει. Εγώ θα σας δώσω κάποιες πολύ προκαταρκτικές σκέψεις Εμείς δεν είχαμε ε, σκεφτεί ενδελεχώς το θέμα του νυχτερινού ε, τερματικού σταθμού, έδινε κάποιες προτάσεις και για τα ενδιαφερόμενα μέρη και ούτω καθεξής. Εγώ θέλω να εστιάσω στα βασικά. Ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές μίλησαν και για κάποια αεροσκάφη πολύ θορυβόδη, τα οποία δημιουργούν ανάλογα υψηλή χορύπανση. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να βρούμε το καλύτερο μέτρο από, σχέση, από ψυχή σχέσης κόστους ωφέλους. Να καθυστερήσουμε την εισαγωγή αυτού του μέτρου, να χάρη όπως πρότεινε το Συμβούλιο. Μήπως όμως τελικά με τον τρόπο αυτό στερούμε από τις αρμόδιες αρχές που θέλουν να μετριάσουν τον θόρυβο ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό οικονομικά μέτρο και συνεχίζει να είναι υψηλή η πίεση για γενικούς λειτουργικούς περιορισμούς οι οποίοι πλήττουν και τις εταιρείε εκείνες που έχουν επενδύσει και επενδύουν σημαντικά ποσά σε πιο αθόρυβα αεροσκάφη. Αυτό είναι το θέμα. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο τέθη από όλους τους ομιλητές είναι το δικαίωμα ελέγχου και η επικουρικότητα. Να επαναλάβω, το έχω πει και στην Επιτροπή Τραν και λέγεται και στο Συμβούλιο, ότι εμείς υποστηρίζουμε πλήρως την εξή λύση. Τα κράτη-μέλη ξεκάθαρα παραμένουν στη θέση του οδηγού και λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις μπορεί να λαμβάνονται από εθνικές αρχές, από δικαστές, από κάποια όργανα ή διαδικασίες διαμεσολάβησης ή οτιδήποτε άλλο. Και εκτιμώ το ότι εσείς έχετε διατυπώσει και κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε όλο αυτό το φάσμα, το εύρος των διαδικασιών. Θέλουμε επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ένα ξεκάθαρο ρόλο, ώστε όλα τα στάδια της διαδικασίας να τηρούνται, να γίνονται με τον σωστό τρόπο. Αν μπορώ να κάνω μια σύγκριση, στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για κανονισμό και όχι για οδηγία, γιατί θέλουμε να ε, δώσουμε μια συνταγή. Αυτά τα βήματα πρέπει να γίνουν για το λειτουργικό περιορισμό κτλ. Αυτή είναι η συνταγή. Θέλετε να φτιάξετε εσείς αυτό το κέικ. Το φτιάχνετε, αν δεν θέλετε δεν το φτιάχνετε, αλλά αυτή είναι η συνταγή. Και η Κομισιόν παρεμβαίνει μόνο αν υπάρχει παραβίαση των σταδίων, των βημάτων της διαδικασίας. Εσείς θα αποφασίσετε αν θα φτιάξετε ή όχι το κέικ. Αν ξεχάσετε να βάλετε ζάχαρη στο γλυκό, θα μπει, θα παρέμβει η Κομισιόν και θα σας πει βάλτε ζάχαρη, γιατί το κέικ δεν είναι καλό. It has nothing to do with the... Αυτό είναι το ζήτημα και δεν έχει να κάνει καθόλου με την ουσία της απόφασης. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το κατά πόσον όλα τα επίπεδα που εσείς θέλετε να δημιουργήσετε για να προστατεύσετε τους πολίτες σας. Δεν έχει να κάνει με αυτά. Μόνο με τη διαδικασία έχει να κάνει. Και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα τώρα να απαντήσω σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σχεση κόστου κόστους-οφέλους και κάποιες παρατηρήσεις ότι δεν ασχολείται με την υγεία η Κομισιόν. Κοιτάξτε, αυτό το θεωρούμε δεδομένο και το ρυθμίζει και η οδηγία περιβαλλοντικού θορύβου, που τα κράτη-μέλη υποχρεώνονται να θέτουν περιβαλλοντικούς στόχους. Εμεί θέλουμε να ενισχύσουμε τη σχέση, τη σύνδεση της εν λόγω οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο και των δράσεων που ε, ενεργοποιούνται, που δρομολογούνται με δυνάμει της οδηγίας αυτής. Και θέλουμε να έχουμε την συνταγή που θα επιτρέπει να λαμβάνονται κατάλληλες δράσεις για τη μείωση του θορύβου. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο κανονισμός είναι το καταλληλότερο νομικό μέσο, διότι ορίζει ξεκάθαρα ποιοι είναι ενδιαφερόμενοι και συμμετέχοντες φορείς. Ορίζει τις, τις και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Αυξάνει τη διαφάνεια για όλους τους ενδιαφερομένους φορείς. Και για τους πολίτες οι οποίοι ζουν κοντά στα αεροδρόμια. Επομένως, η Επιτροπή βασίζεται στην στήριξη της δικής σας Επιτροπής προσβλέπουμε στη συνεργασία και με τον εισηγητή σας αλλά και με όλους εσάς και είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις ενδιαφέρουσες ιδέες που έχετε διατυπώσει που θα ενισχύσουν τη διαδικασία, θα την καταστήσουν πιο διαφανή για όλους όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα και ε, τους επηρεάζει ο θόρυβος, οι χωρί μας αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν και θέλουν όπως είπατε να πάρουν το αεροπλάνο όταν τελειώσει η να γυρίσουν σπίτια τους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τη δυνατότητα στον εισηγητή να απαντήσει σε ερωτήσεις που τέθηκαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο που έχω να κάνω είναι να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου όσους συναδέλφους μίλησαν διότι βλέπω ότι τελικά βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει ένας κορμός όλων των παρεμβάσεων από το οποίο συμφωνούμε. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Η δική μας γνωμοδότηση στην έκθεση της Επιτροπής Αναφορών, της Μεταφορών θα έχει μια διαφορετική εστίαση, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η υγεία και το περιβάλλον. Συμφωνούμε λοιπόν στον κορμό αυτό το γενικό της έκθεσης να ληφθεί υπόψη περιβάλλον υγεία, στην ισορροπημένη προσέγγιση, να διευκρινιστεί ο ρόλος των ενδιαφέρων ε, μέρων και των τοπικών αρχών, το ζήτημα, το ζήτημα του οργάνου διαμεσολάβησης που θα μπορούσε να επιλύει τις διαφορές, τα δικαστήρια και η ισορροπία του ρόλου της Επιτροπής. Αυτά τα θέματα μας ενώνουν και είναι το σημαντικότερο για μένα. Όταν εγώ έθεσα θέμα περί νυχτερινών τερματικών σταθμών, μεταξύ άλλων μέτρων, είπα ότι φυσικά δεν μπορεί να τυποποιηθεί αυτό, γιατί κάπου θα μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το νυχτερινό αεροδρόμιο, αλλά αυτό θα επαληθευτεί επί τόπου, ότι μπορεί ε, να απομακρυνθεί ο θόρυβος ε, με τη μετάθεση κάπου αλλού αυτών των νυχτερινών πτήσεων. Δεν λέω όμως ότι θα πρέπει όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης να έχουν και έναν νυχτερινό τερματικό σταθμό. Επισκέπτομαι πολλά αεροδρόμια, γιατί και ταξιδεύω πολύ, αλλά και ε, πήγα επί τούτου με κάποιου διευθυντέ αεροδρομίου για να μου εξηγήσουν την κατάσταση και μου είπαν ότι δεν γίνεται να γίνει αυτό παντού. Η συζήτηση τώρα περί οδηγία ή κανονισμού. Πρέπει να σα πω ότι ουσιαστικά ήθελα να προκαλέσω, να το συζητήσουμε δηλαδή. Ήθελα να είμαι βέβαιος ότι πραγματικά ε, κάνουμε αυτό που πρέπει και ήθελα να συζητήσουμε όλα τα στοιχεία Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί νομίζω ότι η έκθεση θα είναι πολύ καλή. Και αυτό το αντλώ και από τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την προκειμένη περίπτωση δεν ξέρω, αλλά σε άλλες εκθέσεις που ε, διαχειρίζεται, βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο συνήθως έχει προχωρήσει περισσότερο ε, και τελικά δεν τροποποιείται ιδιαίτερα η θέση μας. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ είναι να συμπεριλάβουμε τις διάφορες απόψεις που ακούγονται και στην τοπική κοινωνία και να προσπαθήσουμε να τις ε, συγκεράσουμε, να τις συμφιλιώσουμε. Τι περιορισμοί πρέπει να εφαρμοστούν. Είναι ένα θέμα, αλλά συζητάμε και κάτι άλλο. Μήπως κάποιοι λειτουργικοί περιορισμοί μπορεί να δημιουργούν περισσότερη χορύπανση. Μιλάμε για λειτουργικούς περιορισμούς σε σχέση με το θόρυβο. Όλα δηλαδή θα περιστρέφονται γύρω από τον θόρυβο. Αν δεν είναι ε, μεγάλος ο θόρυβος που εκπέμπεται από ένα αεροδρόμιο, δεν χρειάζεται να ληφθούν περιορισμοί. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί φαίνεται ότι θα είναι θετική και θα βοηθήσει στην εξέβρεση μιας ε, λύσης που θα οδηγήσει στην καλή αυτή έκθεση. Τώρα αν θα είναι η οδηγία θα δούμε, θα δούμε σε τι συμφωνία θα καταλήξουμε. Αλλά όλα αυτά τα σημεία από των οποίων συμφωνούμε θα περιληφθούν στην έκθεση και κάνουμε και ένα άλμα υπό την έννοια ότι η ενημέρωση, η πληροφόρηση, συμμετοχή των ενδιαφερομένων, τι τεχνολογίε, υγεία, περιβάλλον περιλαμβάνονται. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχο μα. Και έχοντα ακούσει του συναδέλφου, νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο αυτό. Ευχαριστώ όλου και εσά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ την σύνοψη αυτή και πράγματι συχνά η πρόκληση οδηγεί στην ε, ε, ε, παραγωγικότητα. Είχαμε πολύ χρήσιμη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 27 Ιουνίου στις 12. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες στην Επιτροπή μας 19 και 20 Σεπτεμβρίου. 10-11 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Η Επί της, αρμόδιας, ε, ε, επί ουσίας αρμόδια επιτροπή θα ε, ψηφίσει φαίνεται στις 20 Σεπτεμβρίου και το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και περνώ τώρα στο θέμα 19 της ημερησίας διάταξης περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόριξη χιστολιθικού αερίου και πετρελαίου. Η συγητή μα είναι ο συνάδελφος Μπόχουσλαφ Σόνικ. Για λόγους αποτελεσματικότητας, διότι έτσι θέλουμε να λειτουργεί η Ευρώπη, Θα παρακαλούσα τους ε, βουλευτές να φέρουν ε, την επόμενη φορά τις τροπολογίες που βλέπετε ε, εδώ. Πάρτε το μαζί σας και φέρτε το την επόμενη φορά, να μην χρειάζεται να τα ξανατυπώσουμε όλα αυτά. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή. και παρακαλώ όποιον θέλει το λόγο να ζητήσει το λόγο τώρα και όταν ολοκληρώσει ο εισηγητή, ε, θα σας διαβάσω τα ονόματα ε, και θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Ο Μπόξουλαφ Σόνικ, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. 166 τροπολογίε έχουν υποβληθεί στην έκθεσή μου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που καταβάλατε και για την εκπόνηση των τροπολογιών, καθώς επίσης και για τα σχόλιά σας γενικά. Ε, είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν την κεντρική γραμμή της έκθεσής μου, αλλά βεβαίως έχω, υπο... έχω λάβει και κάποιες τροπολογίες οι οποίες ε, θέλουν να σταματήσει εντελώς, να απαγορευτεί η εξόρυξη ιστολιθικού αερίου. Και επίσης ε, ε, να θεωρηθούν ε, σαν απαγορευμένες ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στο υδατικό μείγμα το οποίο χρησιμοποιείται για την, μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα προσπαθήσω να αναφερθώ στις πιο γενικές κεντρικές περιοχές συμβιβασμού. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει όλο και περισσότερο ενεργειακά αυτόνομη και να εξαρτάται όλο και λιγότερο από, την, από εξωτερικούς παράγοντες. Άλλωστε, και στον ενεργειακό οδικό χάρτη ε, για το 2020 αναφέρεται η σημασία αυτού του σχιστολιθικού αερίου στην ανάπτυξη ενός καλύτερου ενεργειακού μείγματος. Βεβαίως θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο η φυστάμενη νομοθεσία και βεβαίως θα πρέπει να βελτιωθεί και η υλοποίησή της εφαρμογή της. Θα πρέπει ε, βεβαίως να υπάρχουν περισσότερες ε, βέλτιστες πρακτικές. Ε, φυσικά θα πρέπει να υπάρξει σωστή επιτήρηση ε, και πρέπει να σας πω και ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας έχει λάβει κάποιες παρόμοιες έτσι, αρχές όσον όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την εξόριξη σχιστολιθικού έργου αερίου. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια σε κάθε επίπεδο και όσον αφορά του εμπλεκόμενους φορεί και όσον αφορά τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Το ίδιο άλλωστε είπαμε ε, στην ε, συζήτηση που είχαμε όσον αφορά τις εξωτερικές ε, εταιρείε μετά από την μόλυνση του Χάτσον. Στην έκθεσή μου αναφέρω και το, τον έλεγχο του μείγματος των υδάτων, την δυνατότητα χρήσης ε, όσο γίνεται λιγότερου ύδατος ε, στη διαδικασία υδραυλικής ρογμάτωσης ε, και επίσης την αφαίρεση κάποιων επικινδύνων συστατικών από αυτό το υδατινό μείγμα. Πιστεύω ότι η εμπειρία που είχαμε μέχρι τώρα σαφώς καταδεικνύει ότι είναι εύκολο να καθησυχαστούν φόβοι. Ε, απ' την άλλη μεριά είναι εύκολο να τρομάξει κανείς τον κόσμο και να παίξει αρνητικά πάνω σε, κάποιες, ε, ε, σε κάποιους προβληματισμούς. Εγώ αναφέρω και στην έκθεσή μου να ε, υπάρχει ότι πρέπει ε, να υπάρξει ενημέρωση του κοινού μέσω εκστρατιών, ευαισθητοποίησης, ε, μέσω ε, πληροφόρησης κτλ. Αλλά βεβαίως αναφέρω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε επιτόπου να υπάρχει και στενή συνεργασία με τις γεωλογικές αρχές και επίσης πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες εξόριξης και η εξόριξη των φρεατίων να υπάρξουν γεωλογικές μελέτες κλπ. Ε, προσπάθησα να λάβω υπόψη τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό σχολείων ε, και νομίζω ότι θα ελβελπιστώ ότι θα φτάσουμε σε συμβιβασμό ε, κυρίως όσον αφορά την χρήση νερού και όσον αφορά και την επιτόπια ανακύκλωση κλειστού βρόχου των υδάτων και την απορροή των χρησιμοποιημένων υδάτων. Ε, στην, στο μείγμα ε, στο μείγμα για, που χρησιμοποιείται για την υδραυλική ρογμάτωση 98 ή 97 περίπου της 100 το λιγότερο είναι, από το μείγμα είναι απλό νερό. 1 έως 3% ε, είναι οι άλλες, τα άλλα συστατικά. Ε, ξαναλέω λοιπόν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες ε, τεχνικές, διαθέσιμες τεχνικές, ότι βεβαίως θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή του ομολύνων πληρώνει και επίσης ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν οι νομοθεσίες που έχουμε, κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον, δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε ε, μελέτη αντικτύπου, ότι θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν και οι εθνικές ε, νομοθεσίες με σωστό τρόπο. Και φυσικά να υπάρχει πλήρης επιτήρηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη συμμόρφωση με τις ε, αρχές ε, ασφαλείας. Μέσα από όλα αυτά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε το σωστό δρόμο για τους ε, συμβιβασμούς και λαμβάνοντας φυσικά υπόψη ότι όλοι ενδιαφερόμαστε για τα πρότυπα υγείας, για τα πρότυπα ασφάλειας οπωσδήποτε, αλλά από την άλλη πλευρά ενδιαφερόμαστε και για την ενεργειακή αυτάρκεια. Θέλουμε επίσης να ε, βελτιώσουμε την κατάσταση και στην Ευρώπη και στον κόσμο όσον αφορά τις εκπομπές ε, αερίων και επομένως ε, θέλουμε ασφαλή ενέργεια που θα μολύνει λιγότερο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Σόνικ για την εισαγωγή αυτή. Προτού να δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές, διαβάζω τα ονόματα. Ρούδι, Judith Merkis, Konrad Simanski und Esther de Lange. Anna Rosbach sehe ich noch. Rosbach. Chris Davis ist Davis. Und wen haben wir? Haben wir dann alle? Αυτά ήταν όλα τα ονόματα. De Rosbach, Davis. Ωραία, κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών και ξεκινάμε τη συζήτηση με τους σκιώδεις εισηγητές. Ελίντα Μακέβαν. Ευχαριστώ. Σήμερα συνεδριάζει για πρώτη φορά η ε, ομάδα των σκιωδών εισηγητών για να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς έχοντας διαβάσει τις τροπολογίες. Κάτι μπορεί να γίνει, αλλά διαφέρουν πάρα πολύ οι απόψεις. Υπάρχουν οι λεγόμενοι, θα έλεγα, cheerleaders που υποστηρίζουν ε, το σχιστολιθικό αέριο και οι εντελώ ε, απολέμοι και κάποιοι που είναι στο ενδιάμεσο. Ε, γενικά υπάρχει και έκκληση να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι είναι μια τεχνολογία την οποία δεν τη γνωρίζουμε καλά και ξέρετε ότι και δεν είναι στη χώρα, παραδείγματος χάρη, κάποια διερευνητική προσπάθεια έχει ξεκινήσει, η οποία δημιούργησε και ε, μικροσυσμούς. Με την εξορρυκτική δραστηριότητα λοιπόν προκλήθηκαν μικροσυσμοί, άρα πρέπει να γίνει ε, πραγματικά μεγάλη μελέτη για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε εξορρυκτικά φρέατια και πόσο ασφαλή είναι αυτά. Αλλά λένε, είναι τόσο παλιά η τεχνολογία που δεν έχει κανένα πρόβλημα, το λέει τροπολογική 21 του κ. Κάλαναν. Όχι, για μια δεκαετία υπάρχει περίπου αυτή η συνδυασμένη τεχνολογία, αν θέλετε. Δεν είναι τόσο παλιά και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Εγώ και τα μέλη της Επιτροπής της ομάδας μου Είχαμε παραστεί σε αυτή την ειδική ακρόαση και μας είπαν ότι η Κομισιόν και διάφορες γάμα δέλτα κάνουν πολύ σοβαρές μελέτες, αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Θα δημοσιευτούν αργότερα φέτος. Μέχρι λοιπόν να έχουμε στα χέρια μας αυτές τις μελέτες, πώς μπορούμε να τοποθετηθούμε για το σχιστολιθικό αέριο. Βέβαια δεν έχουμε αρμοδιότητα να εμποδίσουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν, αλλά νομίζω ότι πρέπει πρώτον να διαβάσουμε τι μελέτε αυτέ, να ακούσουμε τι λένε οι επιστήμονες. Ο κύριος Σόνικ λέει ότι είναι σημαντικό ε, το να είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι και ανεξάρτητοι. Ναι, αλλά δεν είναι ο μόνο τρόπο το λιθικό αέριο, μπορούμε να επενδύσουμε και στι ανανόσιμε πηγέ ενέργεια. Κάτι άλλο εξίσου σημαντικό για μένα είναι οι δεσμεύσει μα ε, για το μετριασμό τη αλλαγή του κλίματο. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μα όταν μιλάμε για νέε ενεργειακέ πηγέ, διότι δεσμευόμαστε από νομικέ απαιτήσει ε, για να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα. Και όποια χώρα ακολουθεί στο μονοπάτι της χρήσης του συστολιθικού ε, αερίου θα πρέπει να τηρεί και κάποιες ε, απαιτήσει για την προστασία του περιβάλλοντος. Για το περιβάλλον, για την ε, ρήπανση των υδάτων πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πρέπει να γίνει βασική έρευνα και για τα επίγεια δεν θα ήθελα δημόσια κονδύλια να πηγαίνουν σε έρευνα για το σχιστολιθικό αέριο προσωπικά, διότι οι εταιρείε αυτέ είναι πάρα πολύ εύρωστε οικονομικά και αν θέλουν να κάνουν έρευνα στην αναλάβουν μόνε του. Και βέβαια και τις χημικές ουσίες πρέπει να ε, προσέξουμε πάρα πολύ. Εκεί ίσως και για το νερό και για τα χημικά καταλήξουμε σε συμβαστικέ προτάσει, για του άλλου τομεί δεν ξέρω. Και κάτι τελευταίο ότι και τα θρακορυχεία ε, προκαλούν προβλήματα για το περιβάλλον, αλλά έχουμε τόσα χρόνια ε, συμβιώσει με ανθρακοριχεία. Και εγώ ζω κοντά σε περιοχή εξόριξης ε, άνθρακα. Σε μας υπάρχει και ένα ταμείο το οποίο πληρώνει για ό,τι πρόβλημα μπορεί να προκύψει από τα ανθρακοριχεία. Ε, ρήπανση, ε, άντληση νερού κτλ. Οι εταιρείε λοιπόν που κερδίζουν τα χρήματα είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να ε, βάλουν και τα κεφάλαια για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων που θα προκύψουν. Ως liability, ως ευθύνη. Στην Πενσιλβάνια έχουν σχιστολιθικό αέριο. Τώρα όμως, δέκα χρόνια αφού ξεκίνησαν, νομοθετούν και μας λένε μην κάνετε το ίδιο. Δηλαδή μας λένε πρώτα νομοθετήστε και μετά ξεκινήστε. Ευχαριστώ η Κορίν Λεπάζ. Ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ακολουθήσω τη γραμμή της Λίντα Μακέβανα να πω εξ αρχής ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες μας ε, που κινητοποιούνται με έντονο τρόπο. Και δεν νομίζω ότι με απλή ε, εκστρατεία ενημέρωση, όπως μας είπε ο κ. Σάντς ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί υπάρχει και πολλή παραπληροφόρηση. Το δεύτερο Οπωσδήποτε θα πρέπει να ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο, το είπε η Λίντα μόλις τώρα. Είναι η δικιά μας ευθύνη να το κάνουμε και είναι κάτι απαραίτητο. Θα πρέπει επίσης να σπάσουμε κάποιες προκαταλήψεις, ας πούμε αυτήν της ε, ενεργειακής ανεξαρτησίας, γιατί θα πρέπει πρώτα να είμαστε σίγουροι για τις ποσότητες που ε, υπάρχουν και δεύτερον ε, να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, για την αυτάρκειά μας. Ε, επίσης, ε, εάν θέλουμε να φύγουμε, να ξεφύγουμε από, τις ορυκτές, από τα ορυκτά καύσιμα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει βεβαίως έτοιμη λύση και η αποτυχία του Ρίο το καταδεικνύει αλλά εάν βάλουμε δημόσια χρήματα ε, στο συστολιθικό αέριο σημαίνει ότι εξακολουθούμε να ε, θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα. Ενίσχυση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πλαισίου. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2011 μετά από παραγγελία της ε, Επιτροπής μας ε, με οδήγησαν σε μια σειρά τροπολογιών σχετικά με την ενίσχυση της νομοθεσίας. Θα ξεκινήσουμε από την εφαρμογή των ε, αρχών της πρόληψης και της ασφάλειας. Πριν από το 2013 θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση της νομοθεσίας σε υφιστάμενους τομείς. Πρώτον, η οδηγία EPPC θα πρέπει και εδώ να βάλουμε την εξόρυξη σχιστολικού αερίου. Δεύτερον, η οδηγία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ε, θα πρέπει να αναφερθούν ε, οι κίνδυνοι της διερεύνησης και της εξόριξης ε, του αερίου αυτού. Τρίτον, στο παράρτημα 3 για την οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης θα πρέπει να προσθεθεί η εξόρυξη αυτού του αερίου. Είναι απαραίτητο επίσης να απαιτήσουμε ε, οικονομικές διασφαλίσεις από τους ε, εμπλεκόμενους έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, οποιοδήποτε ατύχημα σε οποιαδήποτε φάση. Δηλαδή ο εμπλεκόμενος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να, να ε, πληρώσει. Επίσης όσον αφορά τα παράγωγα της υδραυλικής ρογμάτωσης ε, θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να αναφερθούν ε, στην οδηγία περί αποβλήτων ε, και επίσης θα πρέπει να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή πρόληψη όσον αφορά την αποφυγή μόλυνσης. Επίσης το πρόβλημα δεν αφορά το πόσο είναι το ποσοστό των τοξικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ε, στο μείγμα για την υδραυλική ρογμάτωση, αλλά η τοξικότητα των προϊόντων ε, η ίδια. Επίσης, ε, θέλουμε να ξεπεράσουμε τα ορυκτά καύσιμα και όχι μόνο δεν το κάνουμε, αλλά φαίνεται ότι τα αποθέματα αυτού του αερίου δεν είναι και τόσα πολλά όσο θέλουμε. Ε, και μάλιστα η πρόσφατη απόφαση της Πολωνίας ε, από ό,τι φαίνεται είναι ε, λόγω μικρών εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων να μην προχωρήσουν στην εξόριξη. Τώρα θα πω κάτι εξ μου και όχι της ομάδας μου. Εγώ έχω υποβάλει τροπολογία σχετικά με ένα μορατόριο το οποίο θα πρέπει να λάβει χώρα σχετικά με τα προβλήματα τα οποία προκαλούνται από την υδραυλική ρογμάτωση. Προ Προτείνω λοιπόν να υπάρξει ένα μορατόριο όσον αφορά την χρήση της υδραυλικής ε, ρογμάτωσης για την εξόριξη του ε, σχισολιθικού αερίου. Δεν υπάρχει βιασύνη, μπορούμε να περιμένουμε ε, να είμαστε βέβαιοι για την κατεύθυνση προς την οποία θα οδηγηθούμε. Αυτή είναι μια προσωπική τροπολογία, δεν την, έχω υποβάλει εξ της ομάδος μου. Ευχαριστώ πολύ. Η Κορίν η Σαμπίνε Βίλς έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ε, λάθος σειρά. Μισελ Γιβεζή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θέλω να χαιρετήσω τον Σνάλφο Σόνικ, παρότι διαφωνούμε με την εκθεσή του. Γιατί εγώ σκέφτομαι, διαρωτώ με, πού χρησιμεύει αυτή η έκθεση. Κυρίαρχη είναι κάθε χώρα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό τη μείγμα. Και αυτό είναι και φυσιολογικό. Όμως, θα πρέπει η έκθεση παρόλα αυτά να προστατέψει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και θα πρέπει να είναι και συνεπής και συνεκτική με τις επιλογές που ε, γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πακέτο κλίμα ενέργεια. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι Μακάβαν και Λεπάζ διότι πρέπει να μην λέμε τα πάντα και ό,τι να είναι. Συμφωνούμε σε ένα σημείο με τον εισηγητή που λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ε, νομοθεσία για να προστατευθούν τα κράτη από τους κινδύνους που εκπροσωπούν, ε, εκπροσωπεί το σχιστολιθικό αέριο. Και λέει ότι θα πρέπει η εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου να περιληφθεί στο παράρτημα 1 σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είναι άκρος απαραίτητο, γιατί πρέπει να παράγονται πάνω από 500.000 κυβικά μέτρα την ημέρα για να μπαίνει στο παράρτημα. Αλλά ε, με το σχιστολιθικό αέριο μιλάμε μιλάμε για... La deuxième chose. Τεράστιες ε, ε, ποσότητες. Επίσης λέει για την νομοθεσία για τα ύδατα. Η Πολωνία, παραδείγματο χάρη, δεν έχει ποτέ εφαρμόσει σωστά την οδηγία πλαίσιο για τα είδη. Ούτε έχει ένα σύστημα παρακολούθηση ποιότητα ε, των ε, επιφανειακών ε, και, και υπόγειων υδάτων. Πώ θα γίνει λοιπόν με το σχέστο αέρα, αν δεν έχουμε έλεγχο παρακολούθηση και σημαία αναφορά. Και αυτό θα επηρεάσει και την ευθύνη που θα έχουν οι φορεί εκμετάλλευση στη συνέχεια. Και τέλο, όπως υπόθηκε, περιμένουμε πάρα πολλές μελέτες και από την Επιτροπή της ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ Περιβάλλοντος. Δύο μελέτες περιμένουμε για τους υγειονομικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους και για την επίπτωση των περιβάλλων. Εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει πράγματι να υπάρξει μορατόριουμα ε, στην υδρορογμάτωση και την ε, εκμετάλλευση αν δεν δημοσιευτούν πρώτα οι μελέτες και επίσης τηλεφωνήσαμε την Αμερικανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Ε, το πρώτο σχέδιο θα είναι διαθέσιμο στα τέλη του 2012 και το 2014 θα έχουμε όλες τις μελέτες. Υπάρχει καλύτερη από ε, τους από τις που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και που μας λένε μην πιεστείτε και μην βιαστείτε γιατί όταν ε, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Το ξέρουμε αυτό. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι σωστά. Πρώτον, υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ της, ε, του λεγόμενου hydraulic simulation και το hydraulic fracturing. Η υδρορογμάτωση έχει διαφορετική πίεση, ποσότητες νερού και χημικό πρόοδο που χρησιμοποιούνται. Δεύτερον, πακέτο κλίμα-ενέργεια. Εδώ πρέπει να είμαστε συνεπείς με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να λέμε και το βλέπω και στο ΡΕΣΙΝ20. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να μειώσουμε τα αέρα θερμοκηπίου. Έχουν δείξει οι μελέτες ότι η υδρορογμάτωση, επειδή έχουμε έκκληση ε, μελάτων, μετάλλων που επιβαθμίζουν, που ε, υπονομεύουν και αυξάνουν και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, θα μας κάνει να μην μπορούμε να σεβαστούμε τα όρια που έχουμε θέσει. Πώς μπορούμε να ζητήσουμε χρηματοδότηση στο πλαίσιο της έρευνας και της ανάπτυξης για την καλύτερη μέθοδο για την ευρωρογμάτιση. Έχουμε δεσμευτεί να μην μελετήσουμε και να μην χρηματοδοτήσουμε τεχνικές για τα ορυκτά ε, καύσιμα. Άρα θα χρηματοδοτήσουν οι εταιρείε. Τώρα, οι φορείς εκμετάλλευσης λένε ότι υπάρχουν τεράστια αποθέματα ε, και κοιτάσματα. Άρα θα έχουμε ένα ενεργειακό ελντοράντο ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και γεωλόγοι τι λένε, ότι είναι πολύ μικρότερα αυτά τα κοιτάσματα, αυτά τα αποθέματα. Για Exxon Mobil στην Πολωνία θα φύγει από τη χώρα γιατί δεν έχει βρει εμπορικό εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Και κάτι τελευταίο πολύ σημαντικό. Ευθύνη. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μεγαλύτερη νομική ευθύνη για τους φορείς εκμετάλλευσης. Με αυτό το πρόβλημα των εγγύσεων. Διότι και εκεί έχουμε αυτό που έγινε και με τις εκμεταλλεύσεις άνθρακα. Όταν γίνεται υδρορογμάτωση, τι γίνεται, ε, βάζουμε το, το νερό, ε, το υγρό αυτό σε πολύ μεγάλο βάθος που μπορεί τελικά όμως αυτό να μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα που βρίσκεται πολύ πιο ψηλά. Και αυτό να μην γίνει άμεσα, αλλά να γίνει μέσα σε 20-30 χρόνια. Όλοι έχουμε λοιπόν, πρέπει να έχουμε αστική ευθύνη για 20-30-40 χρόνια. Και καλύτερα να γίνει νωρίτερα παρά αργότερα, γιατί μετά ποιος θα το πληρώσει, οι χρήστες και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, θα ήθελα να πω στον εισηγητή ότι πρέπει να γίνει πράγματι μια ισορροπημένη έκθεση. Πρέπει να προστατεύσουμε του Ευρωπαίου πολίτε. Δεν πρέπει να λέμε ότι ναι, ορίστε, θα είμαστε ανεξάρτητοι και τι ωραία που είναι. Εκμετάλλευση στο λιθικό αερίου. Ξέρουμε αν επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα του αέρα, του νοερού και της υγείας και η ανθρώπινη υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κόνρατ Σιμάνσκι στο όνομα του Μάρτιν Κέλεναν. Και έχουμε και μια ομάδα επισκεφτών από την Βαβαρία κατόπιν πρόσκλησης ε, της ε, συνατέρφου Άνια Βάισκερπερ. Καλώς ήρθατε θερμά. Αναφερθήκαμε ήδη στη Βαβαρία ε, σχετικά με τον τρίτο ε, σιδηροδρομικό σταθμό που δεν θα χτιστεί. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα αντικαταστήσω τον συνάδελφο έτσι ώστε να δώσω την επίσημη γνώμη της ε, ομάδας μου για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Τα τελευταία δύο χρόνια άρχισα να δουλεύω ε, στο, για το θέμα ε, των ε, μη, συμβατών, μη συμβατικών συγγνώμη, μορφών ενέργειας. Δεν βρήκα κανέναν ο οποίος θέλει να υποβαθμίσει την νομοθεσία ή τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, θέλουμε να προωθήσουμε, να ενισχύσουμε την νομοθεσία ε, και άκουσα ε, όσους μίλησαν σήμερα ε, και προφανώς οδηγούνται προς την διακατεύθυνση. Κανένας δεν έχει το μονοπόλιο της προστασίας του περιβάλλοντος. Όλοι θέλουμε να το προστατέψουμε, ας πούμε η προστασία των υπογείων υδάτων, του υδροφόρου ορίζοντα η ανακύκλωση ε, του νερού, η χρήση, ε, ε, η δυνατότητα χρήσης των λιμάτων, όλη η διαδικασία επένδυσης, η διαφάνεια των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα τα οποία στηρίζουμε όλοι μας βέβαια. νομίζω ότι τελικά θέλουμε να δουλέψουμε έτσι ώστε να εξευρεθεί μια, ένας κοινός συμβιβασμός που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις ε, ε, θεωρήσεις ε, βλέπω ότι οι τροπολογίες, είναι πολλές. Έχω όμως την εντύπωση ότι δεν είναι όλες επικοδομητικές. Ε, έχω την εντύπωση ότι μερικές είναι λίγο ιδεολειπτικές ε, και ε, επιλέγουν να αγνοούν και την πρακτική των φορέων εκμετάλλευσης αλλά και, τις, και την τεχνογνωσία και τις επιστημονικές αποδείξεις. Ε, νομίζω ότι ε, μου δημιουργείται η αίσθηση ότι γίνεται μία προσπάθεια υποτίμησης ε, αυτού του νέου ορυκτού καυσίμου, να δημιουργηθεί μάλιστα και ένα κλίμα εναντίον αυτού του νέου καυσίμου, το οποίο έδωσε πολλές ελπίδες και προκάλεσε μεγάλη συζήτηση εντός και εκτός της Ευρώπης. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτές τις ιδεολειψίες να επικρατήσουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα ε, στοιχεία ε, κακής ε, πίστης απέναντι στο σχιστολιθικό αέριο και συνήθως ε, αυτά βρίσκονται στα χείλη όσων υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για την μείωση των εκπομπών αερίων ε, του θερμοκηπίου στον πλανήτη μας ε, όμως ε, οι ίδιοι δεν λένε ότι για να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος θα πρέπει ε, να χρησιμοποιηθεί περισσότερο το αέριο στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα καλό σενάριο, η, χρήση, ε, η μεγαλύτερη χρήση αερίου. Και νομίζω ότι από περιβαλλοντική άποψη θα πρέπει να το αναγνωρίζουν και όσοι θέλουν να προστατέψουν το περιβάλλον. Απ' την άλλη πλευρά να μην ξεχνούμε και την οικονομική αξία του αερίου που μπορεί να παίξει σημαντικό οικονομικό ρόλο σε πολλές ε, περιοχές. Αυτή την κατεύθυνση θα ακολουθήσω εγώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το λόγο στη συνάδελφο Βίλς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα αλλά και ήδη στο εργαστήριο συζητήθηκαν ε, πολλοί τεχνικές πτυχές, ε, οι ευκαιρίες και οι ε, κίνδυνοι, ε, αλλά ακούστηκαν ε, επιχειρήματα τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά από τη συζήτηση για την εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας, ότι χρειαζόμαστε το σχιστολιθικό αέριο για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Η η υδραυλική ρογμάτωση αποτελεί γέφυρα προς το πουθενά, διότι μιλάμε για μια παλιά πολιτική η οποία βασίζεται κυρίως ε, στα ορυκτά καύσιμα, καύσιμα και ε, που δεν ε, κοιτάει στο μέλλον. Με την υδραυλική ρογμάτωση θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και τους τελευταίους πόρους που έχει η γη και να τους εκμεταλλευτούμε στο έπακρον θα πρέπει να πληρώσουμε με την υγεία μας, θα πρέπει να πληρώσει η κοινωνία και με ε, ρήπανση των ε, υδάτων ε, και περιβαλλοντική ρήπανση. Η υδραυλική ρογμάτωση υπάρχει εδώ και δεκαετίες, αλλά η μέθοδος, η τεχνολογία και τα χημικά που χρησιμοποιούνται τώρα είναι πιο δυνατά και πιο επικίνδυνα από ό,τι στο παρελθόν. Στόχος είναι να κατακαιρματιστούν λίθινοι όγκοι ε, και αυτό είναι νέο. Βρίσκω απογοητευτικό το σχέδιο του εισηγητή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές. Το δυναμικό του λιθικού αέριου βασίζεται μόνο σε κερδοσκοπικούς υπολογισμούς των ε, ε, εταιριών και στην δική μου χώρα η αρμόδια αρχή ε, υπέβαλε την προηγούμενη εβδομάδα ε, νούμερα τα οποία θα πρέπει να μας κάνουν να το ξανασκεφτούμε. Πολύ μικρό ποσοστό μπορεί πραγματικά, μπορούμε πραγματικά να εκμεταλλευτούμε και επίσης η επιρροή στο κλίμα του, της υδραυλικής ρογμάτωσης είναι χειρότερη από ε, τα συμβατικά καύσιμα. Η Κομισιόν ε, καλείται να ε, χρηματοδοτήσει επιλοτικά προγράμματα, αλλά νομίζω ότι ο τομέας αυτός είναι ο τελευταίος που χρειάζεται ενίσχυση. θα, προσπαθούν να εξοραίσουν τα, τις συνέπειες για το περιβάλλον και για τους ε, κατοίκους ε, στις περιοχές. Πιστεύω ότι θα πρέπει... Γίνεται προσπάθεια επίσης για ε, εκστρατείες ενημέρωσης το κοινού που στόχο έχουν να το καθησυχάσουν. Εδώ και μήνες στη Γερμανία η εταιρεία ExxonMobil ε, διαφημίζει την ε, υδραυλική ρογμάτωση ε, μην χωρίς να αναφέρει τους κινδύνους. Ο κόσμος όμως φοβάται την νέα αυτή τεχνολογία στην περιοχή του. Η έκθεση αυτή είναι απαράδεκτη και μονομερής. Ξανατονίζω, η εκμετάλλευση των ε, μη ε, συμβατών ορυκτών ε, καυσίμων είναι κάτι απαράδεκτο. Με την τεχνική πρόοδο και μόνο δεν είναι δυνατό να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Η τεχνολογική πρόοδος θα πρέπει να συνοδεύεται από αλλαγή στη συμπεριφορά. Και αυτό ιδιαίτερα όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, ε, πολύ μεγάλη πίεση που ασχεί το σχετικό λόμπι εδώ στο Κοινοβούλιο. Βρίσκω ε, αμφισβητήσιμη τη δραστηριότητα του τομέα αυτού. Και θα πρέπει να φροντίσουμε η λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο να γίνεται με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιμάνσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την έκθεση αυτή και να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά του. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας αλλά και έντονη συναισθηματική φόρτιση. κάτι που κατανοώ γιατί το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σημαντικό και για το ενεργειακό μα μέλλον. Κάποιες φορές όμως είναι και δύσκολο να το καταλάβει κανείς, διότι η ίδια η συζήτηση, όπως διεξάγεται, ε, δεν ε, μας δίνει το λόγο να πιστούμε ότι πρέπει ε, να ακούμε και να δεχόμαστε τέτοιες ριζικές και αρνητικές δηλώσεις. Μέχρι στιγμής ο εισηγητής μας, ο κύριος Σόνικ, μας έχει αποδείξει με τη δουλειά του ότι λαμβάνει υπόψη του όλες τις απόψεις και όλους τους φόβους που εκφράζονται. Θέλει όμως να παρουσιάσει και κάποιες νέες δυνατότητες και κάποιες ελπίδες οι οποίες παρουσιάζονται με αυτή την τεχνολογία. Γι' αυτό και με εκπλήσει όταν ακούω ριζοσπαστικές ε, απόψεις ε, όπως αυτή της προηγούμενης συναδέλφου. Νομίζω ότι πρέπει να λέμε ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Και αυτό το επιχείρημα για τα λόμπι μπορούμε να τα αντιστρέψουμε και να μιλήσουμε και για το λόμπι των επιχειρήσεων που είναι κατά αυτών των ορυκτών καυσίμων και που επίσης ασκούν πιέσεις. Καλό θα ήταν ίσως ε, να προσανατολίσουμε τη συζήτησή μας προς τη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά υπάρχουν φόβοι, είναι προφανές και είναι και φυσικό. Όλοι οι πολίτες, ε, όσοι ζουν στην Ευρώπη, φοβούνται. Όπως φοβούνται για τα πυρηνικά ή μπορεί να φοβούνται και για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, φοβούνται για την ρήπανση του νερού. Εύκολο είναι λοιπόν κάποιος να εκμεταλλευτεί το επιχείρημα και έτσι να μπλοκάρει όποια απόφαση προσπαθούμε εδώ να λάβουμε. Καλό θα ήταν λοιπόν να είμαστε πιο ανοιχτοί προς την εξέβρεση μιας συμβιβαστική λύσης. Έρχομαι στις τροπολογίες. Ίσως ορισμένες ε, τροπολογίες ε, να ανάβουν κόκκινο φως, ε, να βγάζουν την κόκκινη κάρτα, ούτε καν κίτρινη κάρτα. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι η τεχνολογία αυτή είναι μια σημαντική εναλλακτική λύση αντί δηλαδή της χρήσης ε, μη καθαρών ε, τεχνολογιών. Η χώρα μου η Πολωνία βασίζεται ε, στον άνθρακα. Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής πολλά. Έχουμε επενδύσει σε χρήμα, σε προσπάθεια. Έχουμε αναστησιστήσει τη χώρα μας μετά την τόση του κομμουνισμού. Τέτοια ριζοσπαστικά σχόλια ε, όταν τα ακούω ε, είναι σαν να μας δείχνουν κόκκινη κάρτα για να είμαι επίκαιρος λόγω του ποδοσφαίρου. Δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό. Η υιοθέτηση πολλών τροπολογιών ουσιαστικά ε, αν γίνει, ε, δεν θα γίνει με συμβιβαστικό πνεύμα και θα καταστρέψει και την δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σόνιτ και νομίζω ότι οι ευκαιρίες ε, θα πρέπει να κερδίζουν, να ε, επικρατούν του φόβου. Δεν θα πρέπει τίποτα να μας υπαγορεύει ο φόβος. Και ουδέτερες εντελώς τεχνολογίες δεν υπάρχουν. Όλες έχουν κάποια αρνητικά αποτελέσματα, ιδίως τα ορυκτά καύσιμα. Το ίδιο πρόβλημα το είχαμε και το συζητήσαμε για τα ορυκτά καύσιμα που είναι στον ε, βυθό της θάλασσας. Είναι αφέλες να πιστεύει κανείς ότι δεν υπάρχει καμία αρνητική επίπτωση. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο και ελπίζω αυτό να μας βοηθήσει και να βοηθήσει την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στους ε, υπόλοιπους ομιλητές. Πρώτα όμως θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά έναν νέο συνάδελφο, Έρικ Πάνκι, από το ΕΛΚ, από την Ουγγαρία. Ήδη έχω μιλήσει γερμανικά μαζί του, με καταλαβαίνει. Ε, καλώς ήρθατε θερμά ως, ε, αναπληρωματικό, ως αναπληρωτής ε, στην Επιτροπή μας. Ε, προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία μαζί σας. Η Ρενάτε Ζόμερ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπόχουσλαβ Σόνικ. Είναι καλή η έκθεση αυτή για ένα πολύ δύσκολο θέμα. Και δεν τη βρίσκω τόσο μονομερή την έκθεση όσο άλλη του Βρίσκω ότι είναι εξαιρετική βάση για να πετύχουμε το συμβιβασμό τον οποίο πάντα επιδιώκουμε στο κοινοβούλιο μας. όσον αφορά την υδραυλική ρογμάτωση, όμως ε, νιώθω ε, και εγώ ένα διχασμό, είμαι και εγώ μηχανικός, ε, είμαι αρκετά ανοιχτή απέναντι σε νέες τεχνολογίες, αλλά με ενδιαφέρει το μεγάλο μέρος του πληθυσμού που θα πρέπει να ασχοληθεί με την υδραυλική ρογμάτωση. Ε, εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ, δεν έχω καμία αντίρρηση ε, όσον αφορά την τεχνική πτυχή, η χημική ε, με ανησυχεί. Και νομίζω ότι αυτή είναι η βασικότερη ανησυχία. Ε, όσον αφορά ε, την δέσμευση του αερίου ε, υπάρχουν τεχνικές. Η Γερμανία έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εξόριξης και εγώ προέρχομαι από περιοχή εξορίξεων αλλά είμαι πολύ επιφυλακτική όσον αφορά την χημική πτυχή της υδραυλικής ρογμάτωσης στην περιοχή μου. Ο Θεός ξέρει ότι έχουμε πολλά προβλήματα παλιά λόγω της εξόριξης ε, και της ε, βιομηχανίας. Η εξόριξη ξεκίνησε πριν 200 ε, χρόνια στην περιοχή μου. Υπάρχουν φρεάτια τα οποία δεν είναι καταχωρημένα. Υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να καταλάβει κανείς διότι παλιά δεν υπήρχε υποχρέωση καταγραφής Υπάρχουν λοιπόν πολλές περιοχές ε, τις οποίες δεν μπορεί να εκμεταλλευτούμε καθόλου ούτε για οικοδομή ούτε για γεωργία. Υπάρχουν ε, περιοχές όπου είναι ε, πάρα πολύ μολυσμένα τα ύδατα. Περιοχές όπου δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος, όπου τα υπόγεια ύδατα είναι μολυσμένα κλπ. Ε, έχει αλλάξει όλη η ροή των υπογείων υδάτων. Επίσης είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε γι' αυτό. Καταλαβαίνω τη θέση ότι σε περιοχές παλαιότερων εξορίξεων δεν θα πρέπει να γίνεται υδραυλική ρογμάτωση. Εμένα με απασχολούν ιδιαίτερα τα υπόγεια ύδατα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι στις ε, περιοχές αυτές ε, δεν ε, λαμβάνουμε το πόσιμο νερό από τα υπόγεια ύδατα, λαμβάνουμε το πόσιμο νερό μας από γειτονικές περιφέρειες. Αλλά οι γειτονικές περιφέρειες στη δική μου είναι ενδιαφέρουσες για τις επιχειρήσεις που θέλουν να εξορίξουν αισχή στο σχιστολιθικό αέριο. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν τις περιοχές μας που έχουν καθαρό νερό για ε, ε, εκμετάλλευση όσον αφορά το σχιστολιθικό αέριο. Προφανώς δεν μπορεί να εγγύθει κανείς ότι ε, τα πολύ τοξικά χημικά θα παραμείνουν στη ζώνη πάνω από τα υπόγεια ύδατα. Αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Το θέμα λοιπόν είναι τι χημικά θα χρησιμοποιηθούν, υπάρχουν επικίνδυνα και λιγότερο επικίνδυνα και φυσικά είναι σημαντικό για την πολιτική και για, τον, ε, για τους πολιτικούς και για τους ανθρώπους, ε, τους πολίτες να γνωρίζουν τι χημικά θα χρησιμοποιούνται και μήπως μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση χημικών, ε, χρειάζονται έρευνες για αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές έρευνες ακόμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε, να μην λάβουμε ακόμα απόφαση, να δούμε ε, τι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα ε, ε μελέτης των ε, διαφόρων γενικών διευθύνσεων ε, της Επιτροπής. Ε, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία δεν μπορούμε να λάβουμε απόφαση. Ε, ας περιμένουμε πόσο μάλλον που τέλος της χρονιάς θα έχουμε τα στοιχεία αυτά. Πιστεύω ότι έτσι θα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο το θέμα αυτό. Ωστόσο πιστεύω και θα πρέπει να τονιστεί αυτό ότι δεν θα πρέπει επί της αρχής να απαγορευτεί το fracking, το, το, το, το, fracking, η υδραυλική ρογμάτωση δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί απέναντι σε νέες τεχνολογίες. Είναι σωστό ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την ε, ασφάλεια ε, ε, παροχής ενέργειας και θα πρέπει να μειώσουμε και την εξάρτησή μας από τρίτες χώρες. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Θέλω λοιπόν πληροφοριακές εκστρατείες ε, καταλαβαίνω το θέμα της, ε, των μελετών ε, των επιπτώσεων στο περιβάλλον και η Λίντα Μακέβαν ήδη είπε ποιος θα πληρώσει μετά. Μπορεί Ε, ο πληθυσμός τελικά να πρέπει να πληρώσει για τις ε, συνέπειες ε, του φράκινγκ της θεραπευτικής ρογμάτωσης μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα, αλλά να φροντίσουμε να είμαστε σίγουροι. Να φροντίσουμε να μην πρέπει οι πολίτες τελικά να πληρώσουν για τις συνέπειες πράξεων που έχουν, που έχουν φέρει κέρδος σε ιδιωτικές εταιρείες. Ιδιαίτερα αν έχουμε ε, εταιρείε από άλλα μέρη του κόσμου θα πρέπει να φροντίσουμε να αναλάβουν την ευθύνη για ενδεχόμενο κόστος που μπορεί να προκύψει μετά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σόμερ. Πρέπει να παρέμβω διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε και μία έκθεση για την αλλιευτική πολιτική στην ημερήσια διάταξη και ο συνάδελφος θα ήθελε να έχει χρόνο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να περιορίσω το χρόνο των επόμενων ομιλητών στο 1,5 λεπτό, αλλιώς δεν θα προλάβουμε καθόλου και έχουν τεθεί πολλές ερωτήσεις προς τον εισηγητή. Θα ήθελα λοιπόν να του δώσω την ευκαιρία να απαντήσει στις ερωτήσεις. Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω, ε, βεβαίω θα προτιμούσα μάλλον, ε, τα όρια να είχαν τεθεί εξ αρχή ε, και όχι τελικά να υποστούν την κύρωση μόνο αυτοί που πήραν τον λόγο τελευταίοι. Εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα που μας απασχολεί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η υδραυλική ρογμάτωση είναι μια τεχνολογία εξαιρετικά επιθετική και επομένως θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ότι πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει γίνει, να έχει ολοκληρωθεί μια πλήρης μελέτη όλων των στοιχείων που θα μπορούσαν ε, να ε, ε, δημιουργήσουν προβλήματα στο παρόν ή στο μέλλον γενικώ δηλαδή μελλοντικά προβλήματα στο υπέδαφος. Πρόκειται λοιπόν για ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Και επίσης ιδιαίτερα προσφυλές ε, μου είναι το εξής, εάν επενδύσουμε σε αυτές τις τεχνολογίες δεν θα έχουμε αρκετούς πόρους για να κάνουμε αυτά που έχουμε ήδη αποφασίσει να κάνουμε, δηλαδή να περάσουμε από τα ορυκτά καύσιμα στα, στις ανανεώσιμες μορφές. Ε, γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε κυρίως την προσοχή μας σε μια ε, σε μια απόφαση κατά την άποψή μου ιδιαίτερα σοφή, την οποία έχουμε ήδη λάβει δηλαδή ε, την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σας ευχαριστώ. Φυσικά έχει δίκιο ο συνάδελφος Βιτόριο Πρόντι ότι ε, ε, έχουμε περιορισμένο χρόνο. Ήθελα να δώσω ε, αρκετό χρόνο στον ε, εισηγητή και τους ε, σκιώδεις και θα έπρεπε φυσικά να έχω περιορίσει και το χρόνο της συναδέρφου Ρενάτε Σόμερ που μίλησε έξι λεπτά. Η συνάδελφος Γιούντιθ Μέρκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πάντα ενδιαφέρον να βλέπει κανείς ε, να διατυπώνονται απόψεις ε, περί πολλαπλότητος ας πούμε των γωνιών από τις οποίες μπορεί κανείς να δει τα επιστημονικά ευρήματα γιατί για μένα η επιστήμη είναι επιστήμη και τα επιστημονικά ευρήματα έχουν μία ε, άποψη. Εν πάση περιπτώσει ακούω εδώ ότι πρέπει να γίνει συμβιβασμός. Μα πώς συμβιβάζεται κανείς με την επιστήμη δηλαδή σε θέματα επιστημονικά πώς μπορεί να επέλθει συμβιβασμός και άλλοι συνάδελφοι πρότειναν ε, να έχουμε πρώτα όλα τα αποτελέσματα των μελετών, όλα τα επιστημονικά στοιχεία από την Κομισιόν πριν πάρουμε απάφαση. Ε, εγώ να σας πω τι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε οτιδήποτε άλλο και να περάσουμε άμεσα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, όσον αφορά τις τεχνολογίες ρογμάτωσης. Ε, νομίζω ότι απλώς ε, δημιουργούμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Στην ουσία ποιο είναι το, το πραγματικό κόστος της υδραυλικής ρογμάτωσης. Ε, λάβαμε υπόψη όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Στις Ηνωμένε Πολιτείες ήδη βλέπουμε ότι λένε ότι 10 χρόνια μετά έχουν πολλά νομοθετικά προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι αν ε, το είχαν σκεφτεί πριν θα είχαν πάρει άλλα μέτρα ε, και προφανώς αυτό που λένε οφείλεται στα κακά αποτελέσματα που είχαν μέχρι τώρα. Το πόσιμο νερό είναι μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να καταλάβουμε ότι ε, ε, περνάει κανείς μέσω της υδραυλικής ρογμάτωσης και πριν φτάσει στην τελική, στο τελικό βάθος περνάει από πάρα πολλούς φλοιούς, περνάει από πάρα πολλά επίπεδα. Έχουμε και τα επιφανειακά ύδατα επομένως τα οποία μπορεί να, μπορούν να επηρεαστούν. Ξέρουμε ότι και στα βαθιά και στα ριχά στρώματα περνάει η ρογμάτωση. Μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ η Άννα Ρόσπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μιλώ εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας. Ε, ε, ε θέλω να κάνω μια δήλωση, διότι μόλις διάβασα ότι η εταιρεία που έκανε εξορίξεις ε, στην Πολωνία ενημέρωσε ότι δεν αξίζει τον κόπο η εκμετάλλευση και γι' αυτό θα σταματήσει. Στη μικρή μου χώρα έχουμε και εμείς αισχύ στο λιθικό αέριο, αλλά η κυβέρνηση πολύ πρόσφατα απαγόρευσε την εκμετάλλευση Συνυπογράφω πρώτον να έχουμε ε, μια σωστή επιστημονική μελέτη των ε, μακροπρόθεσμων ε, προβλημάτων και για, το και για τη φύση και για τα ζώα και για, του, και για τους πολίτες. Θέλουμε δηλαδή μορατόριο πρωτού τα εφαρμόσουμε αυτά. Είχα πάει στην Αλμπέρτα, στον Καναδά και μίλησα με τους ανθρώπους που μένουν εκεί σχετικά με τις ε, μακροπρόθεσμες ε, συνέπειες ε, και τα ζώα τους παθαίνουν λευχαιμία και άνθρωποι αποκτούν ε, καρκινικούς όγκους ε, παρότι οι ε, επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν, ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Επίσης εγώ δει τα δέντρα, ξέρω λίγα πράγματα σχετικά με τα φυτά, εμένα δεν μου φαίνονται πολύ υγιή τα δέντρα και υπάρχουν προβλήματα και για τους πολίτες. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσουμε τους ε, ανθρώπους αυτούς ε, σχετικά με τη ζωή τους. Φοβάμαι ότι κάτι παρόμοιο μπορούμε να πάθουμε και εμείς όσον αφορά το σχιστολιθικό αέριο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Chris Davis, Ο Chris Davis, πράγματι η υδρορογμάτωση είναι πρόσφατη τεχνολογία αλλά 30 χρόνια περίπου παρόλα αυτά ε, η τεχνολογία εξελίσσεται, ιδίω από την πλευρά των ΙΠΑ. Τώρα τα πρότυπα τα περιβαλλοντικά είναι τόσο καλά, αυτό είναι κάτι άλλο. Ε, νομίζω ότι καλά ε, μας ευστά την προσοχή στο θέμα ο κύριος Σεσόνε και υπάρχει αοριστία και ασάφεια σε ό,τι αφορά τεχνολογία και το προς τα που οδεύουμε, δηλαδή σε σχέση με τις εκπομπές, ε, τις εκκλήσεις από την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου. Ε, δεν έχουμε ακόμη ε, μια σαφή απάντηση για το αν ε, είναι μεγαλύτερη σε σχέση με άλλα ορυκτά καύσιμα. Φυσικά και όλοι θέλουμε ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών, αλλά δέχονται όλοι φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει το αέριο που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αν δεν υπάρχει ήλιος, αν δεν φυσάει κτλ. Είμαι αντίθετο στην ιδέα του μορατόριου, δέχομαι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βασιστούμε κάτι που δεν κάνουν ή που δεν έχουν ίσως στην νομοθεσία μας, κάτι που δεν κάνουν οι Αμερικανοί σε σχέση με εμάς. Και έχουμε ένα τελευταίο νομοθέτημα για πρότυπα ε, ποιότητας ε, του περιβάλλοντο και συγκεκριμένα των ε, υδάτων. Επιμένει ότι δεν θα πρέπει επικίνδυνε ουσίες να φτάνουν στα υπόγεια ή στα επιφανειακά ύδατα. Άρα έχουμε την νομοθεσία, απλά πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ πολύ για την ξεκάθαρη σας δήλωση. Κλείνει εδώ κατάλογος των ομιλητών. Δεν μπορώ να πω ότι ζηλεύω τον συνάδελφο Ζόνικ που είναι εισηγητή, γιατί πρέπει να τετραγωνίσει τον κύκλο ουσιαστικά. Θέλουμε ασφάλεια φοδεασμού να έχουμε στον τομέα τη ενέργεια, αλλά Υπάρχουν και πάρα πολλές ε, σκέψεις για την επίπτωση των περιβάλλον. Εγώ για το δικό μου κράτος μέλος πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ε, ε, πολλές πρωτοβουλίες πολιτών, τουλάχιστον έξι. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές από πολίτες για την υδρορογμάτωση και την εξόρυξη στο αερίου άλλες ίσως να είναι προτεραιότητες σε άλλα κράτη-μέλη, άλλες να είναι οικονομικές προτεραιότητες ή προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Σόνικ πάντως για να συνοψίσει, αλλά προηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έχουν τεθεί κάποια ζητήματα που νομίζω ότι σχετίζονται και με την Κομισιόν ή την αφορούν. Παραδείγματο χάρη υποκατάστατα αυτή η μελέτη στις ΕΙΠΑ, για παράδειγμα. Για τα 40-43 εκατομμύρια λίτρα χημικών που αντλούνται, που πηγαίνουν στο έδαφος, αλλά υποτίθεται πρέπει να ε, έρθουν σε επαφή με τον υδροφορορίζοντα. Υπάρχουν επιφυλάξεις από τον τοπικό πληθυσμό, όπως και η κυρία Ζόμερ και εγώ είμαι μηχανικός. Είμαι φίλο τη τεχνολογία, αλλά αυτή η, μέθοδος, αυτή η μεθοδολογία για την εξόριξη σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου είναι λίγο αμφισβητήσιμη. Δεν επαναλαμβάνω, δεν ζηλεύω τον κύριο Σόνικ που πρέπει να τετραγωνεί στον κύκλο. Thank you. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα η εισαγωγή τεχνολογιών όπως είναι η υδρορογμάτωση μπορεί να επιφέρει σημαντικά ωφέλη. Απαιτεί ωστόσο και ιδιαίτερη προσοχή. Και πρέπει να δούμε και τα διάφορα αντισταθμίσματα, το είπαν και πολλοί ομιλητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί ευθύς εξ αρχής να εξασφαλίσει και να σας, να διαβεβαιώσω ότι προσπαθούμε να υιοθετήσουμε μια σαφική και ισορροπημένη προσέγγιση. Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις και φυσικά πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο και εφαρμογή όλων των νομοθετημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να αξιολογεί την ενδεχόμενη ανάγκη ενός πλαισίου αξιολόγησης κινδύνων για το σχιστολιθικό αέριο και εξετάζουμε όλες τις εναλλακτικέ. Η αξιολόγησή μας θα ολοκληρωθεί, όπως αναμένουμε, περί τα τέλη του 2013. Οι, συνεχι... συζητήσεις συνεχίζονται μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως στο πλαίσιο μιας ε, ειδική υπηρεσιακής ομάδας που συμμετέχουν όλες οι υπηρεσίες ε, της Κομισιόν, Ενέργεια, Κλίμα, Δημοσία Υγεία, Επιχειρήσεις κτλ. Νομίζουμε ότι η συντονισμένη προσέγγιση είναι άκρο Επίσης έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών με τα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Είχαμε όμως και πολύ επικοδομητική ανταλλαγή πληροφοριών με τη ΣΥΠΑ. Κάποια από τα σημεία τα οποία έθεσαν ε, οι βουλευτές εμπίπτουν ε, στο πλαίσιο αυτών των συνεχιζόμενων συζητήσεων. Παραδείγματος χάρη, ανάγκη σαφού αναγνώριση και χαρακτηρισμού ορισμένων εργοταξίων ή τοποθεσιών, μέτρηση ποιότητας, ε, ποιότητα νερού και άλλες παράμετρα που πρέπει να μετρήσουμε πριν την υδρορογμάτωση. Επίσης, από τι μελέτες που έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που συνεχίζονται και αναφέρθηκαν από πολλού, θέλω να σας πω ότι μια μελέτη την οποία διενέργησε το ΙΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Περιβάλλον, διενεργεί μάλλον ακόμη, για τον εντοπισμό, την αναγνώριση κινδύνων. Περιμένουμε τα αποτελέσματα να τα έχουμε την δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου. Ε, είναι δηλαδή, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Ελπίζουμε πάντως με τα αποτελέσματα αυτά να στηριχθούν και να, να τεκμηρώσει καλύτερα έτσι τις ε, εργασίες και τις αποφάσεις της η Γενική Διεύθυνση αυτή το Σεπτέμβριο. Τελευταίος ο εισηγητής κύριος Σόνικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους ε, αγαπητοί συνάδελφοι που συμμετείχατε σε αυτήν την πολύ ζωντανή συζήτηση. Μπορούμε να επανέλθουμε βέβαια στο αρχικό ζήτημα. Ε, πρέπει ή δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση. Εγώ πιστεύω ότι ναι, πρέπει να πάρουμε θέση. Έχουμε ήδη πολλές επιστημονικές αναλύσεις. Έχει ήδη παρουσιάσει μία από τις μελέτες η Ευρωπαϊκή, Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, σύμφωνα με την οποία ε, το νομοθετικό υπόβαθρο είναι αρκετό έτσι ώστε να ε, ασχοληθούμε με την νέα αυτή τεχνολογία, ας πούμε, με ασφαλή τρόπο. Ε, τώρα, κάποιες ε, χώρες μέλη έχουν ήδη ε, ξεκινήσει διαδικασίες εκμετάλλευσης της τεχνολογίας. Τα τελευταία 30 χρόνια γίνεται αυτό στην Αμερική βέβαια. Επομένως, προτείνω μια πολύ προσεκτική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τα περιβαλλοντικά στοιχεία θα να βάλουμε δηλαδή μέσα στοιχεία τα οποία σαφώς θα καταδεικνύουν την σοβαρότητα με την οποία να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα. Υπάρχουν βέβαια και συνάδελφοι οι οποίοι λένε ότι η πρόταση δεν πρέπει να, γίνει, δηλαδή ότι θα πρέπει να αρνηθούμε την δυνατότητα αυτής της τεχνολογίας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λογικοί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να δει με πιο ολιστικό τρόπο αυτό το ζήτημα. Αναλύσαμε την ε, νομοθεσία. Βεβαίως θέλουμε να προτείνουμε αλλαγές, αλλά γενικά λέμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε αρκεί να είμαστε προσεκτικοί και σόφρονες. Επίσης να υπάρχει η σωστή ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων, έτσι ώστε οι ντόπιοι πληθυσμοί να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Η προσοχή, η σύνεση πρέπει να είναι πάντοτε ε, το κύριο συστατικό. Και βεβαίως όταν θα έχουμε κι άλλα ε, επιστημονικά στοιχεία, το τέλος του 2013, να επανέλθουμε. Δεν νομίζω ότι το λόμπινγκ της βιομηχανίας είναι τόσο, η άσκηση πίεσης είναι τόσο μεγάλη. Εγώ δεν την αισθάνθηκα τουλάχιστον. Ε, Θυμάμαι ε, ότι όταν ε, η North Stream ε, αποφάσισε να, κάνει lobbying στους υψηλόβαθμους πολιτικούς σε όλη την Ευρώπη είχαν έρθει και σε εμά και είχαμε τότε μία αναφορά και μάλιστα είχαμε και διαδικασία ε, διαδικασία ε, κατά της Επιτροπής έτσι ώστε να αναθεωρηθούν τα περιβαλλοντικά στοιχεία τα οποία συνδέονται με αυτόν τον αγωγό. Λοιπόν, λοιπόν ε, δεν άκουσα τότε φωνές τόσο ισχυρές σαν αυτές που ακούω τώρα. Επομένως, να μην λησμονούμε ότι τα χρήματα τα οποία ενδεχομένως θα εμπλακούν ε, από τα προγράμματα έρευνας για να ελεγχθεί η ε, ασφάλεια της υδραυλικής ρογμάτωσης ε, θα αξίζουν τον κόπο. Ξέρω ότι ήδη υπάρχουν μελέτες έτσι ώστε ε, τα ε, συστατικά που χρησιμοποιούνται στο υγρό για την υδραυλική ρογμάτωση να μην είναι επικίνδυνα. Ούτως ή άλλως δίνουμε χρήματα για, ε, για το καθαρό κάρβουνο, επομένως για το καθαρό άνθρακα, επομένως γιατί να μην επενδύσουμε και σε άλλα τέτοια στοιχεία. Ενδεχομένως το σχιστολιτικό αέριο μπορεί να είναι μία επιλογή και μάλιστα μία πολύ καλή επιλογή. Και βεβαίως εγώ μιλάω από τη δικιά μου πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της χώρας μου και της ε, περιοχής της Ευρώπης στην οποία ε, βρίσκομαι. Όσον αφορά το θέμα της άσκησης πίεσης, το lobbying, το ΕΛΚ έκανε πολλές ακροάσεις ε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα οργάνωσε και εργαστήρια και πραγματικά, πραγματικά ήταν πολλές οι ευκαιρίες που είχαμε να συναντηθούμε και να κάνουμε έτσι μια πολύ ενδελεχή συζήτηση. Ε, ε, είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να συζητήσουμε σε βάθος και σε πλάτος τα ζητήματα αυτά. Να πω κάτι στην κυρία Ρόζεμπαχα. Όταν μιλάμε ας πούμε για τον Καναδά, έχω την αίσθηση ότι ξεχνούμε το πετρέλαιο ας πούμε, το οποίο ε, εξάγεται στο Άλμπερτς από ειδικέ άμμους και νομίζω ότι τότε γίνεται μία προσπάθεια ε, χρήσης μόνο των πολύ επιφανειακών ε, εδαφών. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό όντως μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ε, χλωρίδα και την πανίδα και όντως μπορεί να μην φαίνονται πολύ υγιή τα δέντρα. Ολοκληρώνω. Ο Πρόεδρος είπε ότι το ζήτημα αυτό είναι ε, δύσκολο. Θυμάμαι όταν ήμουνα ε, φοιτητή ε, και αγωνιζόμουν για να ανατραπεί ο κομμουνισμός στην Πολωνία, τότε οι προκλήσεις ήταν πάρα πολλές. Έχω μάθει λοιπόν να αντιμετωπίζω προκλήσεις, δεν έχω πρόβλημα. Ε, γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι σας προτείνω να χτίσουμε μαζί, να οικοδομήσουμε μαζί αυτή την έκθεση, να βρούμε συμβιβασμούς, να σκεφτούμε τους κινδύνους, αλλά βεβαίως να σκεφτούμε και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ε, μιλήσει με καθαρή φωνή σε αυτή τη συζήτηση. Και θα πρέπει να δούμε, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Η νομοθεσία υπάρχει, αλλά ε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον στόχο μας που είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ναι, φυσικά χρειάζεται να καταλήξουμε σε κοινή θέση. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Σήμερα ε, εξετάσαμε τις ε, τροπολογίες ε, στις 19 ε, Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε και προβλέπεται η Ολομέλεια για τον Οκτώβριο του 2012. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα αυτό. Ωραία. Φτάνουμε στο τελευταίο θέμα της ε, ημερήσιας ε, διάταξης για το πρωί. Ευρωπαϊκό Ταμείο της Θαλάσσιας Υποθέσεις και την Αλία. Να δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Χρυσόγελο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν έχουμε επαρκή χρόνο για να γίνει συζήτηση. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι νομίζουν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα ή να μεταθέσουμε τη συζήτηση. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε ε, καλή συζήτηση. Να βρούμε μία λύση ίσως ε, από κοινού. Δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Προτού να ξεκινήσουμε ένα σωρό συζητήσει ε, για τον κανονισμό, ε, προτείνω να ε, ξεκινήσουμε κατευθείαν και να δούμε πόσο θα προλάβουμε. Δέκα λεπτά. Εγώ προτείνω να ξεκινήσετε με την παρουσίαση της νομοδότησής σας και να δούμε πόσο θα προλάβουμε και στο τέλος ε, να δούμε τι θα κάνουμε με τη διαδικασία. Παρακαλώ. τα θέματα της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά για τις παράκτης κοινωνίες και με ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα μια και κατάγουμε από ε, νησιωτική περιφέρεια η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία, που θα αντικαταστήσει το ισχύον Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλία, αποτελεί στοιχείο κλειδί όσον αφορά τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Η κοινή αλληλευτική πολιτική χρειάζεται πράγματι μεταρρύθμιση και το νέο ταμείο πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντο και με στόχο να διασφαλιστεί βιώσιμη αλεία. Η μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτική πολιτική και του χρηματοδοτικού μέσου προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την εξάλληψη των επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην υπεραλίευση, στοχεύοντα τη μετάβαση προ μια πραγματικά βιώσιμη αλληλεία, στην ευημερία των αλληλείων, αλλά και στην επίτευξη υγιών θαλάσσιων οικοστημάτων. Η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία συνδυάζει οικονομικού πόρου για την αλληλεία και τι υδατοκαλλιέργειε, καθώ και για τον έλεγχο και την εφαρμογή των μέτρων, τη συλλογή δεδομένων και την προώθηση ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η ενσωμάτωση αυτών των δύο διαχωρισμένων στο παρελθόν χρηματοδοτικών εργαλείων σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό μέσο μπορεί να απλοποιήσει τη διαδικασία διοίκηση, τη διοίκηση δηλαδή και την ε, διαχείριση μέσω ενοποιημένων κανόνων και διαδικασιών, ενώ θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Η πρόταση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση θα διατίθεται μόνο στα κράτη-μέλη που συμμορφώνονται με τους στόχους και τους κανονισμούς της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και ιδιαίτερα με τις υποχρεώσεις ελέγχου, τον κανονισμό για την παράνομη αλληλεία και τις υποχρεώσεις συλλογής δεδομένων. Επιτρέπει τη χρηματοδότηση των αλληλευτικών επιχειρήσεων μόνο εφόσον συμμορφώνονται με την κοινή αλληλευτική πολιτική. Η πρόταση περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό μέτρων αναγκαίων για να στηριχθεί η βιώσιμη αλληλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα και να βελτιωθούν συνθήκε εργασία μέτρα όπω η προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου, η διευκόλυνση διαφοροποίηση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία, καθώ και η δημιουργία ε, καθώς και η δημιουργία και διαχείριση τοπικών από τα κάτω πρωτοβουλειών για την ενίσχυση τη σωστή βιώσιμη διαχείριση των ελευτικών περιοχών, την προώθηση τοπικών στρατηγικών βιώσιμη ανάπτυξη και των τοπικών συμπράξεων μεταξύ σημαντικών κοινωνικών εταίρων. Προωθεί δηλαδή τη διαβούλευση σε σημαντικό βαθμό. Η πρόταση περιλαμβάνει επίση μέτρα για την υποστήριξη βιοπικιλότητα, συμπεριλαμβανομένη στη διαχείριση αποκατάσταση και παρακολούθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και τη προώθηση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη τη θαλάσσιας βιοπικιλότητα. Τέλο, η πρόταση περιλαμβάνει μερικέ θετικέ διατάξει, οι οποίε θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαφάνεια και την πληροφόρηση του κοινού, να βελτιώσουν τη συλλογή και διαβίβαση δεδομένων καθώ και τον έλεγχο και την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων για την αλεία, παρόλο που δεν ανταποκρίνονται πλήρω σε περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά. Δεν λαμβάνουν υπόψη δηλαδή τι διαφορές που υπάρχουν στι μεθόδου αλεία σε διαφορετικέ περιφέρειε. Ωστόσο, η πρόταση υπολείπεται των προσδοκιών για μια απαραίτητη διαφορετική αλλαγή που θα διασφαλίζει ότι η δημόσια ενίσχυση, δηλαδή η χρηματοδότηση, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προώθηση τη αηφόρου αλείας. Στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία τη διαθέσιμη χρηματοδότηση θα μπορούσε και πάλι να διατεθεί για μέτρα τα οποία ευνοούν μια μερίδα επιχειρήσεων και όχι ολόκληρο τον αλευτικό τομέα ή την κοινωνία γενικότερα. Υπάρχει πολύ περιορισμένη αναφορά στην παράκτεια μικρή κλίμακα αλεία, καθώ και στη στροφή προ μια διαχειριστική προσέγγιση με βάση τα οικοστήματα και την προστασία τη βιοπικιλότητα. Η πρόταση δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τι χρηματοδοτήσει που συμβάλλουν στη διατήρηση τη υφιστάμενη πλεονάζουσα αλευτική ικανότητα, και θα έπρεπε να επιτρέπει τη χρηματοδότηση για πλοία, στόλους και εργαλεία μόνο στη βάση κατάλληλη αξιολόγηση τη αλληλευτική ικανότητα σε σχέση πάντα με τι αλληλευτικέ δυνατότητε, δηλαδή να λαμβάνει υπόψη πόσα ψάρια υπάρχουν σε αλληλευτικά πεδία. Η πρόταση περιλαμβάνει επίση ενισχύσει για τη δημιουργία συστημάτων μεταβιβάσιμων αλληλευτικών παραχωρήσεων, δηλαδή μεταβιβάσιμε άδειε αλληλεία, όταν πολλοί κοινωνικοί φορεί, μη κυβερνητικέ οργανώσει και κράτη-μέλη αντιτίθεται σε κάτι τέτοιο. Κάθε ενίσχυση που αποσκοπεί στη θέσπιση συστημάτων για τη διαχείριση των αλληλευμάτων θα πρέπει να στοχεύει σε διαχειριστικά μέτρα που εμπλέκουν του κοινωνικού φορεί, του κοινωνικού εταίρου σε επίπεδο ελευτικού πεδίου. Η ενίσχυση σκαφών λιμένων για να κάνουν καλύτερη χρήση των ανεπιθύμητων εμπορικών αλληλευμάτων θα υπονομεύσει τι επιθυμητέ υποχρεώσει κατά την εκφόρτωση καθώ και την προσπάθεια να αλλιεύουν πιο στοχευμένα, επιλεκτικά και βιώσιμα ώστε να μειωθούν και οι απορρίψει ψαριών. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να στοχεύει στη μείωση των ποσοστών θνησιμότητα των επιθύμητων αλληλευμάτων, π.χ. μέσω έρευνα για πιο επιλεκτικέ και φιλικέ προ το περιβάλλον πρακτικέ και αλληλευτικά εργαλεία και όχι τόσο στην εμπορία των ανεπιθύμητων αλληλευμάτων. Τέλο, η πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποία θα προωθήσουν αδιακρίτω την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργιών, χωρί την απαραίτητη εξέταση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικέ τροπολογίε που κατέθεσα επικεντρώνονται σε ορισμένα σημεία. Ε, ορισμένοι τύποι χρηματοδότηση, για παράδειγμα, προβλέποντα το σχέδιο, καταργούνται με τι τροπολογίε που κατέθεσα, όπω παράδειγμα ε, για την αποθήκευση ε, ψαριών που αλλιεύονται όταν δεν υπάρχει αγορά. Μεταξύ του να αλλιεύονται ψάρια όταν οι συνθήκε αγορά εγγυώνται καλή τιμή και του να αποθηκεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα τα ψάρια είναι προτιμητέο το πρώτο. Για τα ασφάλιστρα των εκμεταλλεύσεων ιδιωτοκαλλιέργεια, αυτέ οι ενισχύσει δεν είναι λογικέ, με δεδομένο ότι πρόκειται για δαπάνε που πρέπει να επιβαρύνουν του ίδιου επιχειρηματίε και όχι του φορολογούμενου. Επίση, ε, η τροποποίηση αναφέρεται στην, ενίσχυση, στην κατάρριση της ενίσχυσης διαχείριση των, μεταβιβάσεων άδειων, ε, δηλαδή των μεταβιβάσεων αλληλευτικών παραχωρήσεων. Επίση, μια άλλη τροποποίηση αφορά τη διαφήμιση και κυκλοφορία στην αγορά ψαριών για τα οποία υπάρχει περιορισμένη ή καθόλου ζήτηση στην αγορά. Σε αρκετά σημεία προστίθεται διατυπώσει που επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η ενίσχυση, η δημόσια ενίσχυση, δεν έχει ω συνέπεια την υπεραλίευση ή την άκρητη πρόθεση τη Τα κονδύλια ανακατανέμονται για να στηριχθεί η συγκέντρωση επιστημονικών και άλλων στοιχείων και για να βελτιωθεί η επιτήρηση των ελευτικών δραστηριοτήτων. Το τμήμα που αφορά τις υδατοκαλλιέργειε τροποποιείται για να μετατοπιστεί έμφαση προς, από την ε, προαγωγή τη υδατοκαλλιέργεια άνευ κριτηρίων, ενό κλάδου όμω που μπορεί να ε, προξενεί σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα αν δεν τύχει καλή διαχείριση, να, να μετατεθούν οι, οι χρηματοδοτήσεις προς την προαγωγή των δραστηριοτήτων τη υδατοκαλλιέργεια που βασίζονται σε περιβαλλοντικά φιλικότερε συνθήκε. Γι' αυτό η προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τι υδατοκαλλιέργειε δίνεται σε έργα σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνει το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του, δηλαδή να περιορίζονται οι περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Η αλία είναι ουσιαστικά μια ιδιωτική εκμετάλλευση ενό δημόσιου αγαθού, όπω έχει τονίσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και συνοδεύεται κατά συνέπεια από ορισμένε ευθύνε και προποθέσει που περιστρέφονται κυρίω γύρω από τη μέρημνα για αποφυγή τη εξάντληση των αλληλευτικών πόρων ή τη υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντο και των παράθυρων κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτό για την επιβίωσή του. Συνοψίζοντα τέλο, θα ήθελα να πω ότι η χρηματοδότηση πρέπει κατά προτίμηση να αποσκοπεί στη συγκέντρωση δεδομένων που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή αναλύσεων περί βιωσιμότητα των αλληλευτικών δραστηριοτήτων και στη στήριξη όσων ψαρεύουν με τον πλέον βιώσιμο από περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη τρόπο, αλλά και στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της του επικοινότητας μακροχρόνια. Οι τροπολογίες που έχω καταθέσει με την έκθεσή μου είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αποσκοπούν να αδρεώσουν την προσέγγιση ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη μέθοδος, όπως και ότι η βιώσιμη αλληλεία είναι αυτή που βασίζεται σε καλή γνώση και μακροχρόνια διατήρηση του οικοστήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ε, για την εισαγωγή αυτή. Με το μάτι στο ρολόι θα έχουμε τη συζήτηση με τους εσκιώδεις εισηγητές. Το θέμα είναι αν θα το κάνουμε τώρα ή αν θέλουμε να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση στις 3 η ώρα. Ή αν θέλουμε να την έχουμε στο τέλος της ημερησίας διάταξης. Στις 3, ε, Πρόεδρε. Όχι, εγώ δεν θα είμαι και στις 3. Πραγματικά θα πρέπει να περιοριστούμε, διότι και εγώ πρέπει να φύγω. Και έχουμε άλλα θέματα στη μέση διάταξη μετά. 10-15 λεπτά το πολύ θα ήθελα. Να τελειώσουμε και τέταρτο το πολύ. Ούτε καν 15 λεπτά, 10. Ερώτηση προς την Κομισιόν. Η Κομισιόν μπορεί να έρθει στις 3. Βλέπω να γνέφεται καταφατικά. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Thank you,